Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ πολύ. Alors, notre... Λοιπόν, το πρώτο μας θέμα σήμερα είναι η φάρμακο επαγρύπνηση και θα σας πρότεινα να δώσουμε το λόγο λοιπόν στη κυρία Μακάβαν, που είναι η συγγήτρια, για να μας ε, διαφωτίσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα σας δώσω κάποιες ε, πληροφορίες καταρχήν για τους συναδέλφους που δεν έχουν παρακολουθήσει αυτό το φάκελο, ο οποίος είναι αρκετά σύνθετος και μετά θα αναφερθώ σε κάποια πιο εξειδικευμένα θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε και μετά να, ακούσουμε τους Κιώδης και τους άλλους συναδέλφους για άλλα θέματα. Το πρώτο ζήτημα λοιπόν είναι το εξή. Η πρώτη συζήτηση ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί τον Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου. Ε, ζήτησα να μεταφερθεί για σήμερα το πρωί διότι θα έπρεπε να πάω και στην Αγγόλα. Ξέρω ότι αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα διότι αυτό το θέμα είναι ε, μέλος του πακέτου για τα φαρμακευτικά και ε, κάποιοι νομίζουν ότι θέλουμε να το χωρίσουμε. Όχι, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Απλώς ήθελα να γίνει συζήτηση ε, όσο θα είμαι εγώ παρούσα εδώ στην Επιτροπή. Και ε, από την άλλη ενδεχομένως να μην πάω καθόλου στην Αγγόλα τώρα. Εν πάση περιπτώσει εξηγώ στους συναδέλφους ότι θα τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα στην Επιτροπή σχετικά με το πακέτο για τα φαρμακευτικά. Τι είναι η φαρμακοεπαγρύπνηση. Είναι ένα σύστημα παρακολούθησης των φαρμάκων αφού έχουν διατεθεί για δημόσια χρήση. Υπήρξε ένα πολύ σημαντικό τμήμα της δημόσιας υγείας και ξεπλάγει όταν ανακάλυψα από τα στοιχεία της Κομισιόν ότι 5% όλων των ε, νοσοκομιακών ε, συνεπειών είναι από αντιδράσεις από φάρμακα και είναι ο πέμπτος πιο συνήθις θάνατος ε, στα νοσοκομεία προέρχεται από ε, κακή χρήση φαρμάκων. Όταν έχουμε κλινικές δοκιμές, πώς μπορούμε να έχουμε αντιδράσεις, διαρωτάται κανείς, όπως έχουμε και παρενέργειες. Ε, ιδιαίτερα όταν αυτά προκύπτουν μετά από μακρά χρήση ή σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα. Πολλοί θα ε, θυμάστε την ε, τραγωδία τη δεκαετία του 60 των την τραγωδία της Θελιδομίδης τη δεκαετία του 50-60. Συνεπώς χρειαζόμαστε ένα ε, σύστημα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που θα παρακολουθεί τα φάρμακα, θα παρακολουθεί τις συνέπειες και επίσης ε, θα παρακολουθεί τις ε, αντιδράσεις από τα φάρμακα και αυτό αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, η η διαδικασία έχει ως εξής. Η, μια φαρμακευτική εταιρεία υποβάλλει μια αίτηση στο ΕΜΑ και τότε εγκρίνεται ένα φάρμακο. Το δεύτερο είναι με αμοιβαία αναγνώριση, όπου μια χώρα μέλος ε, οδηγείται στην αξιολόγηση ενός φαρμάκου και συντονίζεται με μια άλλη χώρα μέλος για την αμοιβαία αναγνώριση. Δεν, νέα φάρμακα δεν πρέπει να περάσουν από την κεντρική υπηρεσία το, το Συμβούλιο σχετικά με το AIDS και άλλα φάρμακα. Αυτά λοιπόν ε, πρέπει να λάβει κανείς υπόψη, διότι οι κανόνες οι οποίοι διέπουν την συγκεντρωτική υπηρεσία με βάση Ε, με βάση την νομοθεσία 726 του 2004 και το ε, κανονισμό 2183. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει κανείς να αναφέρεται και στις δύο αυτές νομοθεσίες όταν καταθέτει τροπολογίες. Ένα καλό σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης απαιτεί αναφορά των αντιδράσεων από τους ειδικού της εταιρεία και τους ίδιους τους ασθενείς και ένα σωστό συντονισμό από τις δημόσιες αρχές, ούτω ώστε τα διάφορα σημάδια να ανοιχνευθούν. Και μετά θα πρέπει να τα παρακολουθήσει κανείς και να αναλάβει δράση από εταιρείε, δημόσιες αρχές, ούτω ώστε να υπάρξουν τροποποιήσεις στις δόσεις ή στις πληροφορίες που διατίθενται πάνω στο ίδιο το προϊόν ή γενικότερα να ενημερωθεί ο ιατρικός κόσμος. Για πολλά χρόνια είχαμε φάρμακο επαγρύπνηση σε εθνικό επίπεδο και από τη δεκαετία του 90 είχαμε και ένα σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το πλεονέκτημα του ευρωπαϊκού συστήματος είναι ότι δημιουργήσαμε, ε, ε, μια, συγκεντρώσαμε τις πληροφορίες, μια, ένα ευρύ σύνολο πληροφοριών και με αυτόν τον τρόπο η ενημέρωση γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Επίσης, ε, αποφεύγεται η επικάλυψη εργασίας από τις χώρες μέλη για την παρακολούθηση των αντιδράσεων. Έτσι λοιπόν μπορούμε να αλλάξουμε τις πληροφορίες πάνω σε μια ασφαλή φάρμακα πάρα πολύ γρήγορα ο τρόπος με τον οποίο ε, συγκεντρώνονται αυτές οι πληροφορίες, τα σήματα, είναι με αυθόρμητη αναφορά από τους επαγγελματίες την αρμόδια εθνική αρχή, κατά κύριο λόγο, και από τις εκθέσεις ασφαλείας, τις περιοδικές, τα PSUR, τα οποία αναφέρονται και σε πολλές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι εκθέσεις που οι ίδιες οι φαρμακευτικές εταιρείες υποβάλλουν στις δημόσιες αρχές και αναφέρουν ε, αυτά τα οποία έχουν επισημάνει. Επίσης, ε, επίσης πληροφορίες από διάφορα έγγραφα του χώρου, του γιατρικού χώρου ε, και του MEA. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει λοιπόν ένα συντονισμένο σύστημα εδώ και πολλά χρόνια και έχουμε μια ενιαία βάση δεδομένων παγρύπνησης που συγκεντρώνει στοιχεία από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτουργεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο υπάρχουν κάποια κενά στην νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει να καλύψει αυτά τα κενά με την πρόταση που μας υποβάλλει σήμερα. Πολλές από τις ε, πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί είναι καλές ε, πρακτικές, αλλά δεν είναι κωδικοποιημένες και αυτό είναι κάτι το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν τώρα εξετάσει κανείς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, γενικά, εγώ προσωπικά ας πούμε την καλωσορίζω, είναι ευπρόσδεκτη, ωστόσο δεν βλέπω τίποτα επαναστατικό σε αυτήν. Υπάρχουν όμως ορισμένα βασικά σημεία τα οποία θα πρέπει να εξετάσει κάθε βουλευτής. Το πρώτο, μια δομή διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα εργασίας για την επαγρύπνηση. Αυτή η ομάδα εργασίας δεν έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά και υπάρχει γενική συμφωνία από την Κομισιόν, την ΕΜΕΑ e e και από τις χώρες μέλη. Η Κομισιόν λοιπόν προτείνει μια ε, νέα συμβουλευτική επιτροπή αξιολόγησης των κινδύνων για την φαρμακοεπαγρύπνηση και αυτή η συμβουλευτική επιτροπή θα είναι το υπεύθυνο όργανο για την φαρμακοεπαγρύπνηση και θα αναφέρεται στο CHNP που είναι το κεντρικό όργανο που ε, ελέγχει τα ε, φάρμακα στο ευρωπαϊκό σύστημα. Στο Συμβούλιο υπάρχει μια ευρεία συζήτηση σχετικά με την δομή αυτής της νέας Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η Κομισιόν προτείνει ε, να είναι μια επιτροπή γνωμόνων με κάποιους εκπροσώπους από χώρες μέλη, ενώ το Συμβούλιο τίνει προς την κατεύθυνση και επιθυμεί κάθε χώρα μέλος να εκπροσωπείται. Ονομάζεται PRAC, P-R-A-C αυτή η επιτροπή. Η δική μου άποψη είναι ότι ε, πρέπει να παραμείνουμε στην ιδέα του ενός εκπροσώπου από κάθε χώρα μέλος. Η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό θέμα που ενδιαφέρει ε, την κοινή γνώμη. Αν υπάρχει λοιπόν μια απολύτως αντιπροσωπευτική επιτροπή πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο της, ε, να ε, μπορεί δηλαδή να υποβάλει συστάσεις στο CHNP και να έχει αυτή την, αυτές τις αρμοδιότητες. Πολλές αλλαγές ε, προτείνονται ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις αντιδράσεις και συνέπειες. Μια νέα καινοτομία, βασική καινοτομία είναι ότι οι εταιρείε θα πρέπει να αναφέρονται απευθείας στην ευρωεπαγρύπνηση, στο αρμόδιο σώμα αν θέλετε, για κάθε τέτοια αρνητική αντίδραση από φάρμακα. Βλέπω τη λογική αυτού που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αντιλαμβάνομαι επίσης ότι και οι κυβερνήσεις ε, θα ήθελαν να ενημερώνονται πάρα πολύ γρήγορα όταν υπάρχει μια τέτοια αντίδραση στη δική τους χώρα μέλος. Γι' αυτό λοιπόν, α, και στο Συμβούλιο υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην αρμόδια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου επ' αυτού. Πιστεύω ότι πρέπει να, βρούμε κάτι το οποίο θα ικανοποιεί τους πάντες όπου δηλαδή οι εταιρείε να υποβάλουν μία έκθεση στην ε, ευρωεπαγρύπνηση και μετά από τη βάση αυτή δεδομένων της επαγρύπνησης όλες οι χώρες μέλη να ενημερώνονται ε, για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια συμβαστική λύση γύρω από αυτό. Η Κομισιόν επίσης προτείνει όλες οι ε, αντιδράσεις να να αναφέρονται στη βάση δεδομένων της ευρωεπαγρύπνησης από τις αρμόδιες αρχές και τις εταιρείε. Σε κάθε χώρα πρέπει να πω υπάρχει μια αρμόδια υπηρεσία η οποία παρακολουθεί την φάρμακοεπαγρύπνηση, είναι υπεύθυνη για την φάρμακοεπαγρύπνηση σε εθνικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή μόνο σοβαρές αντιδράσεις από φάρμακα αναφέρονται στη βάση δεδομένων της φαρμακοεπαγρύπνησης. Προτείνεται λοιπόν αλλαγή αυτού και να αναφέρονται όλες οι ανεπιθυμητές αντιδράσεις ε, ούτως ώστε να ενημερώνεται η ε, να ενημερώνονται οι περιοδικές ε, εκθέσεις PSUR. Και θα ήθελα να έχω την άποψη των συναδέλφων για το ποιος θα έπρεπε να κάνει αυτή την αναφορά για τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Σε κάποιες χώρες οι ίδιοι ασθενείς μπορούν, έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν ε, στις αρμόδιες αρχές. Αυτό συμβαίνει στη δική μου χώρα εδώ και πολλά χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει όλες οι χώρες να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα, ώστε και οι ασθενείς ως άτομα να μπορούν να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές. Αυτό είναι κάτι που εγώ υποστηρίζω. Ε, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τον ενημερωμένο ασθενή. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν είναι λογικό και λογική αυτή η πρόταση και καλή πρόταση. Άκουσα επιχειρήματα ότι αν επιτρέψουμε και στα άτομα στους ε, επιμέρους ασθενείς να αναφέρουν ε, τέτοιες ανεπιθύμητες αντιδράσεις στις αρμόδιες αρχές, το σύστημα θα δεχθεί υπερβολικά πολλές πληροφορίες και ε, θα υπάρξουν ε, άλλες αντιδράσεις. Εν πάση περιπτώσει, στη βάση δεδομένων τόσο οι εταιρείε όσο και οι χώρες μέλη προς το παρόν τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις ε, δεν μπορούν, δεν μπόρεσαν να τηρήσουν την προθεσμία των 15 ημερών για αναφορά στη βάση δεδομένων. Οι χώρες μέλη είναι χειρότερες. Από πλευράς εταιριών μόνο το 5% καθυστερεί. 50% ε, και πάνω από τις εκθέσεις από τις εθνικές αρχές καθυστερούν πέραν των χρονοδιαγραμμάτων, των προθεσμιών. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη αυστηρότητα, ώστε οι χώρες μέλη να καταθέτουν τις εκθέσεις τους πολύ πιο γρήγορα στην κεντρική βάση δεδομένων. Διότι αν υπάρχουν ανεπιθύμητες ε, αντιδράσεις σε μια χώρα από ένα φάρμακο, πρέπει να το μάθουμε πάρα πολύ γρήγορα, ώστε να ενημερωθούν και οι άλλες χώρες και να εφαρμόσουν ε, ε, τα μέτρα που χρειάζονται. Ένα άλλο ένα, ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό που αποκαλείται IMP, προϊόντα τα οποία παρακολουθούνται εντατικά. Όταν ένα νέο φάρμακο κυκλοφορεί στην αγορά, υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη αυτό το προϊόν να παρακολουθείται και να υπάρχει επαγρύπνηση από αυτού, ώστε να καταγραφούν όλες οι ανεπιθύμητες ε, παρενέργειες, αντιδράσεις. Υπάρχει λοιπόν μια συγκεκριμένη περίοδος παρακολούθησης αυτών των προϊόντων. Αυτή τη στιγμή σε κάποιες χώρες οι ασθενείς γνωρίζουν ότι παίρνουν ένα νέο φάρμακο, διότι πρώτον ο γιατρός τους πρέπει να τους το πει, αυτό δεν συμβαίνει πάντα, αλλά πρέπει ο γιατρός να λέει στον ασθενή ότι παίρνει ένα νέο φάρμακο. Από τη δική μου εμπειρία όμως γνωρίζω ότι οι γιατροί δεν τα λένε πάντα. Κάποιοι μιλάμε και λένε πολλές λεπτομέρειες, άλλοι όχι. Αλλά η Κομισιόν λέει τώρα ότι θα πρέπει μέσα στη συσκευασία του φαρμάκου να υπάρχει κάποια πληροφορία για τον ασθενή, ώστε να γνωρίζει ότι πρόκειται για νέο προϊόν το οποίο βρίσκεται υπό αντατική παρακολούθηση. Α, τούτο υπάρχει, ισχύει σε κάποιες χώρες μέλη. Η Κομισιόν το προτείνει αυτό να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι τούτο θα ενθαρρύνει όλο και περισσότερους ε, ανθρώπους να υποστηρίξουν την προσπάθεια καταγραφής των ανεπιθύμητων αντιδράσεων ADR. Βεβαίως είναι προφανές ότι όλα τα φάρμακα ε, ενέχουν κάποιους κινδύνους. Και θα πρέπει κανείς να αναζητήσει μια ισορροπία. Αν υπάρχουν γιατροί μέσα στην αίθουσα, το μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Όταν οι άνθρωποι παίρνουν φάρμακα, πρέπει να γίνει μια ανάλυση ε, κινδύνων και ωφέλους. Όλο αυτό συνδέεται και με την ε, ιδέα της ε, δυνατότητας για άμεση αναφορά από πλευράς των ασθενών. Υπάρχει μια σειρά προτάσεων για το τι θα πρέπει να συμβεί αν καταγραφεί μια σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση από ένα φάρμακο και τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ενιαίο τρόπο. Στην πρόταση αυτό ονομάζεται κοινοτική διαδικασία, community procedure. Ε, δεν υπάρχει μια τέτοια ενιαία ε, και μοναδική κοινοτική τέτοια διαδικασία και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει. Και ένας άλλος τομέας τελικά είναι η διαφάνεια με την οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις σχετικά με την φαρμακοεπαγρύπνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, ε, η Κομισιόν λοιπόν προτείνει ε, να υπάρχει μια ειδική πύλη στο ΕΜΑ ε, όπου να καταγράφονται όλες οι αποφάσεις και να είναι απολύτως διαφανής αυτή η διαδικασία και μπορεί να υπάρξουν και δημόσιες ακροάσεις ώστε να παρακολουθεί κανείς την όλη διαδικασία. Ε, αυτό είναι παρόμοιο με αυτό που ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Food and Drug Administration. Πρέπει επίσης να πω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που αναφέρεται σε αυτή την μεγάλη βάση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης όπου και οι εταιρείε και οι χώρες μέλη μπορούν να αναφέρουν και να καταγράφονται τα στοιχεία. Αυτή η βάση δεδομένων δεν είναι προσπελάσιμη, ή προσβάσιμη προς τους πολίτες, αλλά η Κομισιόν προτείνει να υπάρχει και μια δημόσια πλευρά ενημέρωσης της κοινή γνώμης. Και αυτή είναι μια εξέλιξη που εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξουμε για να γίνεται ευρύτερη ενημέρωση του κοινού. Αυτά είναι τα βασικά σημεία και εγώ ελπίζω να ολοκληρώσω την έκθεσή μου τις προσεχείς δύο-τρεις εβδομάδες και να τη δώσω για μετάφραση κατά την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Περιμένω λοιπόν να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων επί των προτάσεων αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μακάβαν. Α, συγγνώμη. Είχαμε δει, υποθέτω, και τα δύο θέματα συζητάμε ταυτόχρονα, έτσι, μην τρομάξετε. Το ίδιο και για το 17 και 18. Ε, τα συζητούμε μαζί, είναι κοινή συζήτηση, βεβαίω, λέει η Πρόεδρος, ναι. Ε, ωραία. Η κυρία Πιλάρ Αγιούζο, παρακαλώ σκιώδης εισηγήτρια. Έχετε το λόγο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά την κυρία Μακάβαν για τη δουλειά της. Όχι μόνο επειδή ήταν τόσο επιμελής, αλλά είχε και την καλοσύνη να καλέσει τους σκιώδης ηγητές, να συνεδριάσουμε και να μας τα παρουσιάσει όλα αυτά που σας είπε τώρα εκ των προτέρων. Συμφωνώ σε γενικές γραμμές με όλα όσα είπε. Στο θέμα αυτό δεν θα υπάρξουν πολλές διαφορές μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ε, μερικές λεπτομέρειες ε, μας βρίσκουν σύμφωνους. Είναι πάρα πολύ τεχνικά αυτά τα θέματα, πάρα πολύ περίπλοκα, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία το θέμα και σοβαρά και πολύ ενδιαφέρον θα πρέπει να το εξετάζουμε, πράγμα που κάνουμε κιόλας περιμένουμε την έκθεσή της και όταν θα τη φέρει, αν χρειαστεί, θα κάνουμε και τροπολογίες. Τώρα, για αυτά που είπε η κυρία Μακάβαν επί της ουσίας, για τη δομή του οργάνου λήψης αποφάσεων, αυτό που έχει σημασία είναι ένα αποτελεσματικό. Τώρα, αν συμμετέχει εκπρόσωπος από κάθε χώρα ή δεν συμμετέχει, αν το αποφασίσουν τα κράτη-μέλη, έστω, δεν είναι πρόβλημα αυτό όμως. Το θέμα δεν είναι πόσα μέλη ε, κάθε κράτος μέλος εκπροσωπείται εκεί. Ε, λογικό είναι να θέλει ε, κάθε κράτος να στείλει κάποιον εκεί. Ε, βέβαια, όσο διαφανή και να είναι αυτά και ειλικρινή, είναι λογικό και ανθρώπινο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, είναι να λειτουργεί σωστά. Να είναι καλά και σωστά οργανωμένο, να έχει στηθεί καλά και να δούμε πώς θα λειτουργεί. πώς γίνεται η επικοινωνία και η διαβίβαση των ανεπιθύμητων ενεργειών και αντιδράσεων. Εκεί εγώ κάποια αμφιβολία έχω. Κλονίζομαι λίγο, γιατί δεν είμαι ειδική ούτε σε θέματα κοινή γνώμη, ούτε σε θέματα επικοινωνία και διάδοση. Αλλά μιλάμε για άμεση ενημέρωση, λέτε, από του ασθενεί. Ωραία ακούγεται αυτό. Στο χαρτί ε, γραμμένο καλό φαίνεται για άμεση ενημέρωση, αλλά εκεί πέφτουμε στην υποκειμενικότητα του κάθε ασθενούς Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί ασθενείς που είναι άκρος υποχόνδροι και θα τρομάξουν τον κόσμο. Αφήστε που θα αποπροσανατολίσουν τη δουλειά, θα δώσουν περισσότερο φόρτο εργασίας στους εμπειρογνώμονες. Ο γιατρός λοιπόν πρέπει να το κάνει αυτό. Αν πάρει ένα ασθενή ένα φάρμακο και του προκαλέσει κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ή αντίδραση, ε, να το πει στο γιατρό του. Αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό και ο γιατρός να είναι εκείνος ο οποίος θα βάλει τα στοιχεία στη βάση δεδομένων και θα κάνει την ενημέρωση αυτή. Από την άλλη υπάρχει και άλλος κίνδυνος που είναι υπαρκτός. Να θεωρηθεί ε, εργαλείο και όπλο στον πόλεμο ανταγωνισμού μιας φαρμακευτικής εταιρείας απέναντι σε άλλη. Δεν θα συμβεί αυτό για πρώτη φορά. Το έχουμε ξαναδεί και μπορεί να είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα γιατί θα τσακώνονται μεταξύ τους τα εργαστήρια τα φαρμακευτικά. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ε, και αντιδράσεις συγγνώμη, θα πρέπει να δηλώνονται πολύ νωρίς, τα προϊόντα να παρακολουθούνται ε, εντατικά και θα πρέπει να το ξέρει ο ασθενής αυτό, είτε από το ενημερωτικό σημείωμα μέσα στη συσκευασία, είναι το τοπίο γιατρός ότι κοίτα είναι ένα νέο φάρμακο, ε, τα υπέρ του είναι περισσότερα από τα κατά του, αλλά μπορεί να έχει και σοβαρέ παρενέργειε ή ανεπιθύμητε αντιδράσει, Να το ξέρει αυτό ο ασθενή. Και όταν ανοιχνεύεται ένα περιστατικό που δεν είναι σαφή τα πράγματα, αν οφείλεται το φάρμακο γι' αυτό ή όχι, ε, οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να το γνωρίζουν, να ενημερώνουν και να το θέτουν ε, υπόψη των ενδιαφερομένων πάντα με διαφάνεια. Και σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια τώρα των αποφάσεων και τις δημόσιες ακροάσεις και την ιστοσελίδα και εδώ έχω την ίδια αμφιβολία και θα προτιμούσα να μας το εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, τι εννοείται τώρα να υπάρχει άμεση πληροφόρηση. Η ιδέα της κυρίας Μακάβα να υπάρχει μια ενημέρωση για τους ειδικού και διαφορετική ενημέρωση ε, έτσι πιο εκλαϊκευμένη για το ευρύ κοινό, για τους ασθενείς ή για όποιον ενδιαφέρεται ως καταναλωτής, είναι καλή ιδέα δεν είμαστε όλοι σε θέση να μπορούμε να δεχόμαστε, ε, να επεξεργαζόμαστε και να καταλαβαίνουμε ε, κάθε πληροφορία που απευθύνεται σε ειδικού. Είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχουμε καλές προθέσεις, να τα ε, κάνουμε όλα πολύ καλά και με διαφάνεια, αλλά εδώ κινδυνεύουμε να προκαλέσουμε εμείς παρενέργειες για τη βάση δεδομένων. Βεβαίως να είναι ευρεία για τα φάρμακα χωρίς καμιά αμφιβολία. Συμφωνώ. Δεν θα πρέπει για όλα τα θέματα να έχει την ίδια ένταση, την ίδια πυκνότητα η πληροφόρηση. Ακόμα και σε χρονικά διαστήματα μπορεί αυτό να διαφέρει. Τι άλλο έχουμε. Να, τη βάση δεδομένων το είπα. Δημόσιες ακροάσεις. Ναι, Και εδώ έχω τις ίδιες αμφιβολίες με την άμεση ε, δημόσια ενημέρωση. Α, κάτι άλλο που θα ήθελα να σας πω. Τα φάρμακα κοινόχρηστης ονομασίας, ε, generics, ε, είναι φάρμακα που θα πρέπει και αυτά να υπόκεινται στην ίδια διαδικασία με τα, τα υπόλοιπα που προστατεύονται από εύρυση τεχνίες. Μπορεί να μην είναι νέα φάρμακα και που να είναι σε έντονη παρακολούθηση, αλλά θα πρέπει και για τα φάρμακα αυτά να υπάρχουν στοιχεία. Γιατί είναι φάρμακα που σε πολλές χώρες ακόμα δεν έχουν μπει στο σύστημα και δεν γίνεται ευρύτερη κατανάλωση. Αν ξέρει ο καταναλωτής ή ο ασθενής ότι αυτό το φάρμακο παρακολουθείται λιγότερο ας πούμε στη φαρμακοεπαγρύπνηση θα έχει ακόμα μεγαλύτερη επιφύλαξη ή δισταγμό να το πάρει. Είναι υπέρ των φαρμάκων λοιπόν κοινόχρηση τη ονομασία αυτό να ξέρει ο ασθενή ότι υπόκειται τον ίδιο έλεγχο, την ίδια, ε, στον ίδιο έλεγχο και εφίσταται την ίδια επαγρύπνηση και τα παρακολουθούμε, όχι ότι είναι δεύτερη κατηγορία φάρμακα α πούμε. Καλό θα ήταν η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα τα εξηγήσει όλα αυτά. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα, Η Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία Ριβαζή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα της οδηγίας για τη φαρμακοεπαγρύπνηση, γιατί είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Έχουμε αυτό το θέμα της γρήπης, το πρόβλημα της γρήπης ή τα 1 ή 1 και ανάλογα με τις χώρες, τα πάντα εξαρτώνται από την επαγρύπνηση των αρχών για τη μελέτη των παρενεργειών. Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Τι η Σουηδία ένα εκατομμύριο έχουν εμβολιάσει ήδη στη Σουηδία. Τέσσερις μέρες μετά είχαμε τέσσερις νεκρούς. Και έγινε χαμός. Και τώρα ψάχνουν να βρουν από τι πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι. Από το εμβόλιο ή όχι. Και 194 περιπτώσεις είχαμε με ανεπιθύμητες ενέργειες και αντιδράσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δανειστούμε αυτό το παράδειγμα, να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και αν υπάρχει αρκετή ενημέρωση για τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Γιατί να δούμε το ιστορικό. Κοιτάξτε τι έγινε με το βιόξ. Καρδιαγκιακά ε, επεισόδια θανατηφόρα, κυκλοφόρησε το φάρμακο το 1999 και αποσύρθηκε το 2004. Πέντε χρόνια δηλαδή κράτησε η κυκλοφορία. Ε, κάτι δεν πάει καλά τότε. Αν δούμε το Προζάκ, που αύξησε το ποσοστό αυτοκτονιών. Το ίδιο, δηλαδή από τη στιγμή που κυκλοφορεί και δίνεται η άδεια, υπάρχει καθυστέρηση μέχρι να αποσυρθεί, ακόμα και αν έχουμε δει τι παρενέργειε. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη σε αυτή την οδηγία, θα πρέπει να αναλύσουμε πάρα πολύ καλά πώ λειτουργεί για να βελτιώσουμε το σύστημα. Κυρία Μακάβαν, κάνατε προτάσει που εμπλουτίζουν το κείμενο ε, των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω μερικά ερωτηματικά εγώ. Ερωτηματικό πρώτο τι γίνεται με τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου. Τι είναι αυτό το σχέδιο. Είναι δυνατότητα που έχει ε, ένα νέο φάρμακο να περιορίσει τις άδειες κυκλοφορίας και να αυξήσει την επαγρύπνηση. Καλώς. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά θα πρέπει πραγματικά να είναι η εξαίρεση, διότι μπορεί να είναι ακριβώς κίνδυνος κάτι τέτοιο για να κυκλοφορούν νωρί οι άδειε ε, και τα φάρμακα να βγαίνουν νωρί στην αγορά. Μετά, διαχείριση δεδομένων. Σε ορισμένα κράτη μπορούν άμεσα όντω οι ασθενείς να ε, κοινοποιούν τις παρενέργειες και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Σε άλλες χώρες μεσολαβεί το υγειονομικό προσωπικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η κοινοποίηση, όντως, γιατί ο ασθενή γενικά πηγαίνει στο γιατρό του και του λέει ότι είχα τι τάδε παρενέργειε και ανεπιθύμητε αντιδράσει. Και ο γιατρό τα εισάγει σε ένα σύστημα αυτό, σε μία έκθεση και το δίνει στις αρμόδιες αρχές, στην επαγρύπνηση, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάπου θα πρέπει να υπάρχει μία διήθηση, ένα φίλτρο των στοιχείων αυτών. Ε, δεν έχω πρόβλημα να τα λένε οι ασθενεί, αλλά για να είμαστε αποτελεσματικοί, να ξέρουμε πολύ συγκεκριμένα πώ θα διαβιβάζονται αυτά τα στοιχεία για να αντιμετωπίζονται. Και η πρόσβαση. Εκπλήσουμε πάρα πολύ που οι περιοδικές εκθέσεις ασφαλείας, ενημερωμένε δηλαδή, είναι ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά τα φαρμακευτικά εργαστήρια και κανέναν άλλον. Οποιοδήποτε εξωτερικό αποκλείεται. Υποτίθεται ότι είναι η εμπιστευτικότητα ή το εμπορικό απόρριτο. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι δημόσια αυτά τα έγγραφα. Η μέγα βάση δεδομένων ε, για την επαγρύπνηση. Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να έχουν ε, πρόσβαση, λέει, οι αρμόδιες αρχές της κάθε χώρας. Και ρωτώ, αν εγώ είμαι ένα σωματείο, μία ένωση και έχω έναν εμπειρογνώμονα που θέλει να κοιτάξει το τάδε φάρμακο κοινόχρησης ονομασία ή όχι, τι παρενέργειε έχει και τι ανεπιθύμητε αντιδράσει, θα πρέπει να ζητήσει την άδεια τη αρμόδια αρχή για να έχει πρόσβαση. Μα πώς θα γίνει έτσι η ευρύτερη επαγρύπνηση. Όλοι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβαση. Έρχομαι τώρα στη χρηματοδότηση, άλλο πρόβλημα. Τερματίζεται η υποχρέωση δημόσιας χρηματοδότησης και αυτό απειλεί το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης σε κάθε χώρα. Δηλαδή, παροχή υπηρεσιών είναι αυτή των φαρμακευτικών εταιριών. Εδώ θέλει να είμαστε εμείς προσεκτικοί και να επαγρυπνούμε. Οι παρενέργειες θα πρέπει να κοινοποιούνται και στις εταιρείε αλλά και στις αρμόδιες αρχές. Γιατί η εταιρεία μπορεί να το κρύψει αυτό, να το μπλοκάρει. Από κάπου δεν θα πρέπει να δημοσιευθεί όταν υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι θα το στείλουμε στην ίδια την εταιρεία. Αυτά σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν και άλλα σχόλια αλλά αυτό το θέμα της νέας γρήπης θα πρέπει να μας χρησιμεύσει ως παράδειγμα να δούμε σε κάθε χώρα πώς διαβιβάζονται οι προφορίες. Στη Γαλλία, ας πούμε, έχουμε πρόβλημα. Οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν, αλλά δεν το κάνουν, να δηλώνουν. Στα νοσοκομεία, για παράδειγμα, υπάρχει ένας ιατρός αναφοράς που συγκεντρώνει όλες αυτές τις παρενέργειες και σε αυτόν απευθύνονται. Αυτός είναι ο φύλακας, ας πούμε, που πρέπει να επαγρυπνεί. Φανταστείτε τώρα ε, πόσο, πόση όρεξη έχουν οι γιατροί να το κάνουν αυτό και μετά οι πυρογνώμονες ανεξάρτητοι που θα πρέπει να το ελέγξουν ε, που δεν έχουν σχέση με τα φαρμακευτικά εργαστήρια και τις εταιρείες να δουν λοιπόν αν ευθύνεται για τους θανάτους το εμβόλιο ή όχι. Και πολύ γρήγορα να γίνονται όλα αυτά. Και ε, επαναλαμβάνω όχι μόνο οι φαρμακευτικές εταιρείε. Και σας λέω ενημερωτικά ότι όταν κάναμε την ερώτηση στη ε, Σουηδία στα φαρμακευτικά εργαστήρια η απάντηση ήταν ότι ναι, είχε ε, περισσότερη νέα ενεργή, άλλη ενεργούση, αυτό που λέγεται adjuvant, ε, γιατί με διαφορετικό τρόπο κυκλοφορεί το εμβόλιο σε κάθε χώρα. Το εμβόλιο της GlaxoSmithKline απαγορεύεται στις εγγύους και στα παιδιά στη Σουηδία. Πάτε σε άλλη χώρα και σας λένε όχι, μα αυτό πρέπει να το δώσετε το εμβόλιο στους εγγύους και στα παιδιά. Φλουαρτιστικ δηλαδή, χαιρετίσματα. Ο κόσμος αντί να ξέρει τι γίνεται ε, οδηγείται σε μεγαλύτερη σύγχυση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η οδηγία. Ε, θα πρέπει να έχουμε ε, μεγάλες ιδέες και να, να μην έχουν τόσα πολλά δικαιώματα οι εταιρείε ώστε να βγάζουν πολύ γρήγορα και πολύ νωρί τα φάρμακα στην αγορά, να εθαρρύνονται οι ε, κρατικές αρχές ε, να έχουν δικούς τους εμπειρογνώμονες και διαφάνεια και η κοινοποίηση να είναι σωστή και με καλό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ριβαζή. Θα μιλήσω κι εγώ Τώρα εξ ονόματος της κυρίας Παρβάνοβα η οποία είναι και σκιώδης συζητής της ομάδας μας. Και ειδού αυτά που ήθελε να πει. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πρόσδεκτη ε, με την έννοια ότι έχει ως στόχο να εξορθολογήσει το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης στην Ευρώπη. Πρόκειται ε, για μια προσπάθεια το, το σύστημα να γίνει αποτελεσματικό, διαφανές, ε, πρόληψη, ε, σύστημα πρόληψης. Έτσι λοιπόν ε, με γοργότερο τρόπο θα ε, καταγράφονται οι ε, παρενέργειες και οι ανεπιθύμινες αντιδράσεις προς όφελος του κοινού. Η συζήτηση θα πρέπει να καταλήξει σε ένα σύστημα το οποίο θα εγγυάται ότι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα του συστήματος φορμακοεπαγρύπνησης στην Ευρώπη με στόχο να εγγυάται στο υψηλότερο επίπεδο την ασφάλεια του ασθενούς. Το να μιλάει κανείς για τα φάρμακα μιλάει για τα ωφέλη των φαρμάκων αλλά και τους κινδύνους. Από γιατρική άποψη αυτές οι δύο έννοιες είναι αλληλένδετες και πρέπει να τις έχουμε υπόψη όταν συζητούμε που έχει σχέση με τη φύση της μεταχείρισης των φαρμάκων. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η συμπεριφορά του ασθενή απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους τους κινδύνους από τη χρήση φαρμάκων. Η διαφάνεια, η ενημέρωση, η πληροφόρηση σχετικά με την φαρμακοεπαγρύπνηση θα θα εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή και είναι προς το συμφέρον και του ασθενούς αλλά και των επαγγελματιών υγείας και της βιομηχανίας στην οποία θα πρέπει να έχει εμπιστοσύνη ο ασθενής. Με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η πρόταση μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πρόσδεκτη, διότι ενισχύει την Τράπεζα Δεδομένων Φαρμακοεπαγρύπνησης, κάποια όμως σημεία θα πρέπει να εμβαθυνθούν. Η ενημέρωση των ανεπιθύμητων ε, παρενεργειών που παρατηρούνται με την ε, ενημέρωση από τον ίδιο τον ασθενή. Ε, με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ο ιδιωτικός χαρακτήρας των στοιχείων που συγκεντρώνονται ε, για την τράπεζα δεδομένων και να μπορούν αυτά να χρησιμοποιούνται από άλλους ενδιαφερομένους. Ο ρόλος των επαγγελματιών βεβαίως δεν θα πρέπει ε, να ξεχαστεί. Πάντοτε όταν υποβάλλονται οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Ε, η επεξεργασία θα πρέπει να γίνεται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και θα πρέπει να ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει θέσει στην ε, αγορά το φάρμακο κάθε φορά που υπάρχει τέτοια καταγγελία από τον ασθενή ή τον επαγγελματία. Σχετικά με την ενημέρωση των ασθενών, πρέπει να είμαστε απολύτω σαφείς. Καταρχήν εδώ μιλούμε για μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης. Συνεπώς δεν χρειάζεται να ανοίξουμε νέα συζήτηση για την ενημέρωση των ασθενών. Θα πρέπει να είναι αξιόπιστες, κατανοητές και αντικειμενικές οι πληροφορίες που δίνονται στον ασθενή. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να αναφέρω ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι βασικές πληροφορίες, οι παρατηρούμενες ανεπιθύμενες ενέργειες και να συμβάλλουν στην κατανόηση των πληροφοριών αυτών για τον ε, ασθενή πάνω στην ε, στο ίδιο το φάρμακο. Αυτό είναι προ όφελο του ασθενή και τη θεραπεία του. Τέλο, ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και κάποια άλλα θέματα στη συζήτηση. Η περιοδική έκθεση ασφαλεία, ποια έγγραφα πρέπει να είναι να δημοσιοποιούνται και υπό ποια μορφή, ενώ η νέα επιστημονική επιτροπή που θα επιφορτιστεί με τη φαρμακοεπαγρύπνηση θα πρέπει να είναι σαφής ο ρόλος της, η δράση της, αν θα είναι δημόσια ή μη δημόσια. Απαιτείται λοιπόν μια ευρύτερη συζήτηση όπου σε κάθε φάση οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι στο σύστημα θα εκφέρουν την άποψή τους. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε στη συζήτησή μας ότι η ενίσχυση του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης δεν θα πρέπει να αποτελέσει περιορισμό αλλά πρόοδο για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη του ασθενούς. Ιδού λοιπόν εξ ονόματο της κυρίας Παρβάνοβα. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Westlund. <coughs> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν ήθελα να, να αναφερθώ στον εμβολιασμό και την γρήπη των χείρων. Αλλά επειδή αναφέρθηκε το θέμα, νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ε, από ό,τι ξέρω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ε, πέθαναν δύο άτομα λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό. Ήταν άτομα ε, βαριά άρρωστα και κανένας γιατρός δεν σκέφτηκε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στον εμβολιασμό και τον θάνατό τους, διότι ήταν βαριά ασθενείς. Ωστόσο, είναι καλό το ότι έχουμε μια τέτοια ανοιχτή διαδικασία και ότι παίρνουμε σοβαρά τέτοιου τύπου μηνύματα. Ωστόσο, οι πολύ περισσότεροι έχουν πεθάνει στη χώρα μου από τη γρήπη των χείρων. Άνθρωποι που ε, ήρθαν σε επαφή με το σύστημα υγείας, ε, θεωρήθηκε ότι δεν χρειάζονται τίποτα και μετά ε, πέθαναν μεταξύ άλλων τρία παιδιά Ε, μάλλον ένα παιδί το οποίο ήρθε σε επαφή με το σύστημα υγείας τρεις φορές προτού να πεθάνει στην εντατική. Στην, ε, Φιλανδή, στη Φιλανδία ένα κορίτσι είχε βήχα και πέθανε την ίδια, την ίδια νύχτα και διαπιστώθηκε ότι πέθανε από τη γρήπη των χείρων. Σημαντικό είναι να μπορεί να λάβει κανείς περίθαλψη όταν πάθει γρήπη των χείρων. Χιλιάδες άνθρωποι ε, νιώθουν ότι χρειάζονται γιατρική περίθαλψη, ε, τους θέλουν όμως σπίτι, δεν τους ε, δέχονται στα ιατρικά κέντρα. διότι για τη γρήπη πρέπει να λάβει κανείς γιατρική περίθαλψη μέσα σε 8 ώρες. Κανένα γιατρικό κέντρο όμως δεν αναλαμβάνει τόσο βραχυπρόθεσμα ασθενείς. Υπάρχει εδώ μια πτυχή που αφορά το περιβάλλον, ε, διότι τα φάρμακα επηρεάζουν πολύ το περιβάλλον και σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να αποφύγουμε τις αρνητικές συνέπειες. Ε, στη χώρα μου η ε, βιομηχανία φαρμάκων είναι πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική και έχουν καταβληθεί προσπάθειες για να αποφευθούν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον. Θα θέλαμε στην ομοθεσία αυτή να συμπεριληφθεί το ότι θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη πώς επηρεάζει ε, ένα φάρμακο όχι μόνο την υγεία του ασθενούς αλλά και τη δημόσια υγεία γενικά και το περιβάλλον. Ε, ξέρω ότι στην ε, Σουηδία υπήρχε κάποια υποστήριξη για το νομοθέτημα αυτό. Και ε, είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει και τις αρχές ε, που ασχολούνται με την ε, έγκριση των φαρμάκων. Το θέμα των συνεπειών στο περιβάλλον δεν θα, δεν θα πρέπει ποτέ να επηρεάσει την ασφάλεια του ασθενούς. Εάν όμως υπάρχει φάρμακο που έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, θα πρέπει ο παραγωγός ε, να έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει τις συνέπειες στο περιβάλλον ή να μην εγκριθεί ένα φάρμακο εφόσον υπάρχουν ε, άλλα παρόμοια τα οποία όμως δεν έχουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον. Ή φάρμακα που έχουν ε, εγκριθεί και εν συνεχεία φάνηκε ότι έχουν αρνητικέ συνέπειε για το περιβάλλον θα πρέπει να παρακολουθούνται και θα πρέπει να εξετάζεται μήπω υπάρχουν καλύτερε αναλλακτικέ λύσει. Το θέμα, δεν, το θέμα στο κάτω-κάτω είναι η υγεία των ανθρώπων, διότι το πόσιμο νερό είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο. Και το πίνουν και έγκυες και παιδιά και, το, και γενικά οι άνθρωποι Θα πρέπει λοιπόν ο ασθενή να δικαιούται το καλύτερο δυνατό φάρμακο. Τούτου λεχθέντο όμω υπάρχει λόγο η παραγωγή και να ερευνήσουν ε, τις συνέπειες για το περιβάλλον, αλλά και θα πρέπει να μην εγκρίνονται φάρμακα τα οποία είναι μεν καλά για τον ασθενή, που ε, να έχουν ε, όμως πολύ σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον, εφόσον υπάρχουν καλύτερες αλλακτικές λύσεις. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν αυτές οι δύο πτυχές στην νομοθεσία αυτή. Νομίζω ότι ε, είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον, καθότι ε, τα φάρμακα είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα όσον αφορά τη δημόσια υγεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Πέτερ Λίζε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Λίντα Μακάβαν για την καλή εισαγωγή της. Ε, γενικά συμφωνώ μαζί της. Η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι πράγματι πολύ σημαντικό θέμα. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα διαπιστώνονται οι, ε, κάποιες παρενέργειες. Ε, για να ε, λάβουμε υπόψη μας ε, αυτό το θέμα λοιπόν θα διαρκεί ακόμα περισσότερο και θα στοιχίζει πολύ περισσότερο η έγκριση ενός νέου φαρμάκου. Θα πρέπει να δούμε το θέμα υπό το σωστό φως. Οι ασθενεί που παίρνουν φάρμακα είναι άρρωστοι. Όσο πιο άρρωστοι είναι, τόσο πιο δραστικά θα πρέπει να είναι τα φάρμακα, άρα να έχουν και ε, ε, σοβαρότερες παρενέργειες. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει όγκο, παίρνει, λαμβάνει χημειοθεραπεία. που έχει πολλές αρνητικές ε, συνέπειες και στα λευκά και στα αριθρά αιμοσφαίρια. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι είναι λάθος να κάνει κανείς ε, χημειοθεραπεία, διότι ε, πιο πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνο παρά από τις παρενέργειες της χημειοθεραπεία. Κάποιοι μπορεί, σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να είναι υπερβολική χημειοθεραπεία, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η χημειοθεραπεία από μόνη τη είναι λάθο. Θα πρέπει αυτό να το έχουμε κατά νου. Κάποιες παρενέργειες όμως μπορεί να, είναι, μπορεί να μπορούν να αποφευθούν εάν ε, είμαστε πιο προσεκτικοί. Και φτάνω στο επίμαχο θέμα της πληροφόρησης των ασθενών. Εάν δεν προσέξουμε και εξετάσουμε με κριτικό μάτι την πρόταση του κυρίου Φερχόγεν, τότε μπορεί κάλλιστα οι πληροφορίες των επιχειρήσεων προς τους ασθενείς να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη χρήση νέων φαρμάκων από ό,τι μέχρι τώρα. Αυτό το κατέστησε σαφές η Λίντα ε, ε στα νέα φάρμακα είναι πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος ε, παρενεργειών επειδή δεν υπάρχουν ε, χρόνια πείρας με τη χρήση τους. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στην ενημέρωση και στην διαφήμιση, Ε, θα, ε, μπορεί αυτό να ενέχει κινδύνους, ε, θα πρέπει να... Διότι μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή εισοδήματος σε ένα νέο φάρμακο. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να ξαναεξεταστεί η πτυχή αυτή, ώστε να μην δημιουργούμε κίνητρα για έμεση διαφήμιση νέων και όχι απόλυτα γνωστών φαρμάκων πολύ συγκεκριμένα για την πρόταση αυτή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην απαραίτητη ενίσχυση της φαρμακοεπαγρύπνησης και στην υπερβολική γραφειοκρατία. Θα ήθελα να θίξω εδώ δύο θέματα. Καταρχήν τα PSURs, Δεν θα πρέπει να έχουμε εδώ υπερβολικές απαιτήσεις, διότι θα οδηγήσει σε αυξημένο φόρτο, ιδιαίτερα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το όφελο για την ασφάλεια των φαρμάκων μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ισορροπημένη θέση. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά την σχετική φιλολογία από τις έρευνες. Ε, ο μεγαλύτερος φόρτος ε, για τις εθνικές ε, αρχές και τις επιχειρήσεις σίγουρα δεν θα συμβάλλει στην καλύτερη νομοθεσία. Η πείρα μου μου δείχνει ότι κάποιοι ασθενείς είναι πολύ καλά ενημερωμένοι, ιδιαίτερα όσον αφορά ασπάνιες ασθένειες. Υπάρχουν ασθενείς που μερικές φορές γνωρίζουν καλύτερα την ε, ασθένειά τους και τις ε, θεραπείες από τον μέσο γιατρό. Η πείρα μου εμένα μου δείχνει ότι πολλοί ασθενείς πιστεύουν ε, ότι έχουν παρενέργειες από τα φάρμακα. Μετά από μια συνομιλία με τον γιατρό διαπιστώνεται ότι αυτά είναι συμπτώματα της ασθένειας και όχι παρενέργειες. Μπορεί δηλαδή να μην πρόκειται για παρενέργειες, μπορεί να πρόκειται για κάποια μόλυνση, για κάποια ασθένεια. Ε, σε περίπτωση που διαπιστώσει ο γιατρός κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται να το αναφέρει. Διότι έτσι ούτε παίρνουμε σοβαρά την επιστήμη, ούτε έχουμε κερδίσει τίποτα σαν αφορά το φάρμακο. Τέλος, η Κομισιόν πρότεινε στο σημείωμα που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία να συμπεριληφθεί κεφάλαιο που να λέγεται ε, σημαντικές πληροφορίες. Χθες το βράδυ, ε, σε μια εκδήλωση της, ε, μιας ένωσης της φαρμακοβιομηχα... Ε, φαρμακευτικής βιομηχανίας συζητήθηκε το θέμα του μαύρου πλαισίου και θεωρήθηκε ότι αυτό είναι σαν να είναι ε, ανακοίνωση κηδείας. Αν μας ενοχλεί το μαύρο, είπανε κάποιοι, μπορούμε να το κάνουμε ροζ γαλάζιο, αλλά δεν είναι αυτό το αποφασιστικό ερώτημα. Το αποφασιστικό θέμα είναι εάν έχει νόημα μέσα στη συσκευασία να υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να διαβάσει ούτω ή άλλω ο ασθενή και να είναι γραμμένο με μεγαλύτερα γράμματα. Εγώ νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι λογικό. Χθε σε άλλη συζήτηση άκουσα ότι οι αρχές έγκρισης πιστεύουν ότι το σημείο που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία θα πρέπει να ε, ότι είναι ε, κατανοητά. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι, απλά, ότι είναι ε, ευλήπτα. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες τι οποίες δεν χρειάζεται καθόλου ο ασθενής. Ε, ο παραγωγός όμως για νομικού λόγους είναι υποχρεωμένος να τα ε, γράψει όλα αυτά, αλλά αυτό δεν βοηθάει κανέναν. Στην ε, έκθεση της Λίντα Μακάβαν ή του Κρίστοφ Φιέλνερ θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την πρόταση αυτή, πιστεύω να υπάρχει δηλαδή ένα τμήμα στο σημείο μας της συσκευασία, ε, το οποίο να ε, είναι ξεκάθαρο με μεγάλα γράμματα, εύληπτο, ε, όχι απαραίτητα με μαύρο πλαίσιο για να μοιάζει με ανακοίνωση κηδείας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται εκεί οι σοβαρότερες, οι σημαντικότερες πληροφορίες διότι αυτό που αυτή τη στιγμή συμπεριλαμβάνεται στο σημείωμα της συσκευασία ε, μπορεί από νομικής άποψης να είναι απαραίτητο, αλλά δεν βοηθάει πάρα πολύ τους ασθενείς. Θα πρέπει να εργαστούμε πάνω στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πέτερ Λίζε. Ποιος ε, είπε ότι είναι τα σημειώματα δυσανάγνωστα. Ε, ο Βιτόριο Πρόντι τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το αντικείμενο αυτό της φαρμακοεπαγρύπνησης και πιστεύω ότι είναι σκόπιμο πραγματικά να αφιερώσουμε αυτό το χρόνο και ιδιαίτερη προσοχή. Καταρχά, θα ήθελα να πω ότι κάθε φάρμακο συνοδεύεται από ένα ενημερωτικό σημείωμα και αυτό ενδεχομένως ε, μπορεί να έχει και ε, υποδείξεις για ενημέρωση. Πώς ε, πρέπει να λαμβάνεται να προσλαμβα... και επίσης στα διάφορα στοιχεία μπορούμε να δίνουμε και το όνομα του γιατρού που συνταγογράφησε το φάρμακο αυτό για να φτάνουμε στην πηγή της ενημέρωσης. Διότι θα πρέπει τα στοιχεία αυτά να είναι χρήσιμα και ε, τελικά οι δηλώσεις για τις παρενέργειες και τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις να συλλέγονται με τρόπο ε, ομοιογενή και να έχουν και ένα συγκεκριμένο στόχο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πολύ σημαντικό να έχουμε μέθοδο. Ε, τι εννοώ, ε, και να ξέρουμε το στόχο μας. Ε, τα νέα φάρμακα για να κυκλοφορήσουν στην αγορά χρειάζονται μια διαδικασία, μια έγκριση και μια άδεια. Και από τη στιγμή που κυκλοφορούν, πολύ γρήγορα πρέπει να έχουμε και τις απαντήσεις και τις αντιδράσεις των ασθενών για να ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται το φάρμακο αυτό. Όλα αυτά γίνονται ήδη στη φαρμακοεπαγρύπνηση από τη στιγμή που κυκλοφορεί ένα φάρμακο στην αγορά. Ωστόσο, υπάρχει και ένα πρόβλημα που συνδέεται με τους διάφορους χρήστες των φαρμάκων. Θα ήθελα να θυμίσω ένα κίνδυνο Ξέρετε ότι ορισμένοι ρηπαντές μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές στο νοσοποιητικό σύστημα ε, και σε αλλεργίες. Έχουμε και φαρμακογενείς αλλεργίες. Ε, και εδώ είναι πολύ σημαντικό το θέμα της φαρμακοεπαγρύπνησης. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τα φάρμακα, να ξέρουμε τι προκαλούν ε, στους ασθενείς και πώς αντιδρά το ανοσοποιητικό σύστημα κάθε φορά. Γιατί τα φαινόμενα είναι όλο και πιο συχνά. Και έχουμε και αλληλεπιδράσεις φαρμάκων μεταξύ τους. Αυτέ λοιπόν οι κλιματικές αλλαγέ, τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά μπορούν να προκαλέσουν τέτοια τροποποίηση του ανοσιοποιητικού συστήματος ε, του ασθενούς ε, που να αντιδρά διαφορετικά στην πρόσληψη του φαρμάκου. Αυτά είναι τεχνικά θέματα βέβαια, αλλά θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να αξιολογούν τα στοιχεία για να καταλήγουμε στα σωστά αποτελέσματα. Ο κύριος Ρώση. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό το επιχείρημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ε, ευαίσθητο το θέμα. Και καλό είναι ε, να συνεργαστούμε. Ε, συμφωνώ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τους συναδέλφους. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό να βελτιωθεί το σύστημα φαρμακό επαγρύπνησης, αλλά μην έχει επιπλέον κόστος έμεσο ή άμεσο για τους ασθενείς. Και ε, ε, ούτε για τις εταιρείες που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αν έχουμε επιπλέον φόρτο οικονομικό θα υπάρχει πρόβλημα με την κατάσταση. Θα φύγουν οι εταιρείε. Το 5% των εσόδων ε, των εισαγωγών μάλλον στα νοσοκομεία οφείλεται σε ανεπιθύμητες ε, αντιδράσεις και παρενέργειες φαρμάκων. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι οι ασθενείς να δηλώνουν ε, τα προβλήματά τους στους γιατρούς, σε κάποιον που να έχει γνώση και να είναι ειδικό. Δεν μπορεί ο κάθε ασθενή να γνωρίζει όλα αυτά που χρειάζονται ε, όπως ο οικογενειακό γιατρό ή ένας γιατρό ε, νοσοκομιακό, για να τα βάλει στο σύστημα και να ενημερώσει. Επίσης δεν είναι όλα τα φάρμακα τα ίδια. Α πούμε, ένα φάρμακο είναι αλλεργιογόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Αλλά για πολλούς άλλους ε, ασθενεί, να είναι καλό το φάρμακο δεν μπορεί να κινδυνεύσει να σταματήσει η κυκλοφορία του και να απαγορευτεί επειδή υπήρχαν κάποιες αλλεργίες χωρίς να έχει κυκλοφορήσει άλλο υποκατάστατο. Υπάρχουν λεγόμενες ε, σπάνιες ασθένειες και τα ορφανά φάρμακα ε, που δεν ε, έχουν υποκατάστατα ή εναλλακτική ουσία, εναλλακτικό φάρμακο. Αν υπάρχει λοιπόν ένα μοναδικό φάρμακο για μία αρρώστια και κυκλοφορεί στην αγορά και έχει παρενέργειες, ε, δεν θα πρέπει να το απαγορεύσουν και να μην υπάρχει κανένα φάρμακο για την αρρώστια αυτή μετά. Επειδή με μονομένες περιπτώσεις εμφάνισαν αλλεργίες, που καμιά φορά μπορεί να είναι και κατά φαντασία, να μην οφείλεται το φάρμακο για αυτές, δεν θα πρέπει λοιπόν να απαγορεύεται μετά η συνταγογράφηση φαρμάκων που είναι χρήσιμα και ε, υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν απόλυτη ανάγκη. Σας είπα για τις εταιρείε ε, και να μην επιβαρυνθούν επιβολικά και το ενημερωτικό σημείωμα που συνοδεύει το φάρμακο θα πρέπει να είναι εύληπτο με πολύ συγκεκριμένες στοχευμένες πληροφορίες. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολύ συχνά οι ασθενείς τι κάνουν. Αγοράζουν το φάρμακο, πετάνε τη συσκευασία όπως είναι μαζί με το σημείωμα και μετά έχουν το φάρμακο στο φαρμακείο τους χρόνια ολόκληρα, τα χάπια, τα σιρόπια, ξέρω εγώ τι, μπορεί να έχουν λήξει και όλα αυτά και παίρνουν λιγμένα φάρμακα. Θα πρέπει λοιπόν τα πιο σημαντικά στοιχεία να αναγράφονται πάνω στο φάρμακο, πάνω στο φιαλίδιο ας πούμε και όχι στη συσκευασία ή στο σημείωμα γιατί αυτά μπορεί κανείς να τα πετάξει πολύ συχνά τα κράτη-μέλη και η ίδια μου η χώρα, η Ιταλία δηλαδή, δεν ασχολούνται με το θέμα αυτό. Ας πούμε, υπάρχει ένα πρόβλημα με ένα εμβόλιο, με ανεπιθυμητές ενέργειες ή με αντιδράσεις, οι αλλεργίες, οτιδήποτε. Πολλές φορές δεν ασχολούνται οι χώρες και καλό είναι να ασχοληθεί η με αντιδρασεις αλλεργιες οτιδηποτε πολλες φορες δεν ασχολουνται οι Ένωση για να δραστηριοποιούνται και οι αρμόδιοι οργανισμοί σε κάθε χώρα. Και να αποζημιωθούν οι ασθενείς. Τώρα, τι γίνεται με τα φάρμακα που εισάγουμε από τρίτες χώρες. Βεβαίως γίνονται ε, έλεγχοι των δραστικών ε, ουσιών, αλλά θα πρέπει να δούμε και τη γραμμή παραγωγής τους. Πώς παράγονται, ποια είναι η διαδικασία. Ο κύριος Πρόντι Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα του περιβάλλοντος. Μπορεί να μην έχουν την κατάλληλη δραστική ουσία ή την κατάλληλη ποσότητα. και τι κατάλοιπα. Καμιά φορά μπορεί να περιέχουν και κατάλοιπα ε, τα φάρμακα μέσα λόγω της ρήπανσης και να έχουμε αλλεργίες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και συσκευασίες light. Άλλο πρόβλημα στις συσκευασίες. Ας πούμε, τα χάπια, ε, τα δισκία, να είναι πιο μικρές οι συσκευασίες. Αν κάποιος πρέπει να πάρει 8 χάπια, γιατί να είναι υποχρεωμένος να αγοράσει ένα κουτί που έχει μέσα 16 ή 20 γιατί αυτό τον ε, ενθαρρύνει να ε, συνεχίσει να το τελειώσει το κουτί ε, για να μην το πετάξει και να παίρνει φάρμακα άσκοπα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα πειράματα σε ζώα. Σε λίγο καιρό θα συζητήσουμε αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας για τον περιορισμό των δοκιμών σε πειραματόζωα και τελικά την απογόρευσή τους. Ε, λοιπόν, θέλουμε πραγματική φαρμακό επαγρύπνηση και ενεργητική. Δεν, θα, δεν, επιτρέπεται να δεχόμαστε να κυκλοφορούν φάρμακα που δεν έχουν ε, δοκιμαστεί, που δεν έχουν γίνει πειράματα αρκετά. Σε πειραματόζω, τι να κάνουμε. Λυπάμαι κι εγώ πάρα πολύ. Ε, δεν θέλω να βασανίζονται τα ζώα, αλλά δεν μπορεί να κυκλοφορεί ένα φάρμακο και να πεθαίνει ο κόσμος, ε, οι άνθρωποι δηλαδή χωρίς να έχει δοκιμαστεί το φάρμακο. Αν χρειάζεται πειραματόζω, πειραματόζω. Τι να κάνουμε. Άλλη παρατήρηση. Για τις δραστικές ουσίες. Γνωρίζουμε ότι στη φαρμακοποιία υπάρχουν ενεργές δραστικές ουσίες που επιτρέπονται για διάφορες ομάδες του πληθυσμού. Παράδειγμα, μια δραστική ουσία, ένα ενεργό συστατικό που δεν προκαλεί προβλήματα στους Ευρωπαίους μπορεί να προκαλέσει τεράστια προβλήματα αν χορηγηθεί σε άλλη ομάδα πληθυσμό, ενώ άλλης γεωγραφικής προέλευσης. Στην Ευρώπη όμως τώρα ε, ζουν πολλοί άνθρωποι από όλα τα έθνη, από όλους τους λαούς. Γι' αυτό σας παρακαλώ να γράφει η ετικέτα ε, του φαρμάκου ποιες είναι οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις και οι παρενέργειες για τις διάφορες ε, εθνικές ομάδες. Αφήστε δε που περισσότερες φορές ε, οι άνθρωποι αυτοί δεν μιλούν τη ε, γλώσσα της χώρας και τη γλώσσα στην οποία αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες στη συσκευασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ και να αναγράφονται όλα αυτά στα αγγλικά. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων, τη βιοδιαθεσιμότητά τους και να υπάρχει και ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ε, συναγερμού σε περίπτωση που ε, έχουμε ένα πρόβλημα σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διακοπεί η κυκλοφορία ή για να απαγορευτεί ενδεχομένως να έχουμε κάποια παρέμβαση. Θα πρέπει να εναρμονίσουμε τους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ανάβω και το ρολόι, αλλά δεν βλέπω να έχει κανένα αποτέλεσμα. Ο κύριος Τρεμόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούγονται και για τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Θα ήθελα να συνεχίσω όμως τις ε, σκέψεις που κατέθεσε η κυρία Ριβάση. Και καλό να το δούμε και εμείς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο συνολικά το ζήτημα από την πλευρά των πολιτών και όχι της φαρμακοβιομηχανίας. Ακριβώς γιατί πέρα από τα κέρδη τους βλέπουν, μόνο την καταπολέμηση του συμπτώματος και όχι την αντιμετώπιση της αιτίας όπως μας ε, καλούσε εδώ και κάποιες χιλιάδες χρόνια ο Ιπποκράτης. Βεβαίως και μιλάμε για δυνατότητα αναφοράς των πολιτών σε περίπτωση που υπάρχει καμενής επίδραση στην υγεία του από τα φάρμακα. Αρκεί βέβαια να ζει. Ήδη ακούσαμε από την κυρία Μακάβαν ότι ο πέμπτος πιο συνήθις θάνατος στα νοσοκομεία προέρχεται από τα φάρμακα. Που σημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις, πέρα από τις ιατρογενείς ασθένειες, υπάρχουν και επιπτώσεις σοβαρές από την ίδια την χρήση και όχι την κατάχρηση των ε, φαρμάκων. Χρειάζεται μια ουσιαστική, ουσιαστική και πλήρης πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία και αυτό είναι δεδομένο. Το επιχείρημα που ακούσαμε ότι μπορεί να εμπλακούν σε αυτού του είδους τη διακίνηση πληροφορίας και εταιρείε για λόγους ανταγωνισμού με διασπορά ψευδών ειδήσεων κλπ. κλπ. Δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να το κάνουν και τώρα, αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν γίνεται. Ακριβώς γιατί φαίνεται να υπάρχει και μια προσπάθεια συγκάλυψης αυτών των αρνητικών επιπτώσεων και γι' αυτό οι πολίτες που ψάχνουν να βρουν τι πραγματικά συμβαίνει ή, ε, βρίσκουν κάποιες από τις ε, μελέτες που γίνονται, λίγες σε σχέση με ένα τόσο σοβαρό θέμα, ή διακινούν την πληροφορία μέσα από το ίντερνετ. Τελικά αναρωτιέμαι μήπως κάποιοι φοβούνται ότι αυτή η πρόσβαση πλήρης των πολιτών στην πληροφορία θα σημαίνει και την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων όπου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και δικαστικά για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων. Βεβαίως και ο φορέας φαρμακοεπαγρύπνησης που συζητούμε θα πρέπει να έχει πραγματική δύναμη και αρμοδιότητες. Από την άλλη όμως δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια αποδυνάμωση της διαδικασίας ελέγχου και επιστοποίησης των φαρμάκων πριν την αδειοδότηση. Αυτό μπορεί να σημαίνει στην πράξη ότι θα μετατραπούμε όλοι μας σε ένα μεγάλο πεδίο ερευνητικό, δηλαδή σε ζώντα πειραματόζωα. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει αυτό το σημείο να το προσέξουμε ιδιαίτερα και κλείνω λέγοντας ότι σαν συνέχεια αυτής της σκέψης ότι πρέπει εμείς να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της υγείας ως βασικού αγαθού ατομικού και συλλογικού από την πλευρά των πολιτών και όχι της φαρμακοβιομηχανίας ότι θα πρέπει το ζήτημα αυτό των φαρμάκων, της επαγρύπνησης πάνω σε αυτά να μεταφερθεί από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων στη Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ζιλ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά πάσα πιθανότητα με το φάκελο αυτό, με το θέμα αυτό, αλλά επίσης και με τον κανονισμό και την οδηγία που συζητήσαμε τον Μάιο και είμαι ο, ο σκιώδης για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρόκληση λοιπόν στην Ευρώπη, σχετικά στην Ευρώπη τον 21ο αιώνα. Ε, γενικότερα για τους Ευρωπαίους. Και όλο και πιο στεναρά είναι τα ερωτήματα τα οποία τίθενται. Πολύ συχνά ε, οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται τα φάρμακα τα οποία καλούνται να ε, λάβουν. Και μπράβο στη Λίντα Μακέβαν για τις προτάσεις και για την εισήγηση που μας έκανε στην αρχή της συζήτησης αυτής. Θεωρώ ότι μια οδηγία και ένας κανονισμός για την φάρμακο επαγρύπνηση όχι μόνο θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε το σύστημα, αλλά θα βελτιωθεί και η ενημέρωση του κοινού της κοινή γνώμης και θα υπάρξουν και οι απαραίτητοι μηχανισμοί για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν ε, για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και η βεβαιότητα του ασθενούς στα φάρμακα τα οποία καλείται να πάρει. Παραδείγματο χάρη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το εμβόλιο για τη νέα γρήπη, τα 1 e ένα. Στη Γαλλία, παραδείγματο χάρη, ο εμβολιασμό θα αρχίσει στις 12 Νοεμβρίου. Όσοι δεν επιθυμούν να κάνουν το εμβόλιο μάλλον αυτοί οι οποίοι δεν επιθυμούν να κάνουν το εμβόλιο είναι πάρα πολλοί, ακριβώς επειδή δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι ε, όπως ακριβώς ε, θα έπρεπε να είναι ενημερωμένοι όπως περιγράψαμε σήμερα. Τούτο σημαίνει ότι μια οδηγία όπως αυτή, ένας κανονισμός, είναι εξίσου σημαντικός στην εφαρμογή του όπως ακριβώς και η καταπολέμηση της γρήπης ήταν ένα, ή ένα αυτή τη στιγμή με την ε, χρήση ενός εμβολίου. Δεύτερον, ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι το ζήτημα της επιτήρησης των φαρμάκων. Το ανέφερε και η Λίντα Μακέβαν. Ένα βασικό δεδομένο το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι μόνο το 5% των προβλημάτων που προκύπτουν διοχετεύονται στο κεντρικό σημείο ενημέρωση στη βάση δεδομένων. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο ανταγωνισμός. Ένας ανταγωνισμός μεταξύ των φαρμακευτικών εργαστηρίων και να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η υπέρταση. Πρόκειται για μια ασθένεια όπου υπάρχουν αρκετά φάρμακα. Οι ασθενείς καλούνται να κάνουν χρήση αυτών των φαρμάκων επί σειράν ετών. Κάποιος ισχυρίζεται ότι το δικό του φάρμακο είναι καλύτερο από κάποιο άλλο και ε, το φάρμακο αυτό χρησιμοποιείται μεταξύ 15-20 ε, χιλιάδων ε, ασθενών. Το πώς θα γίνει η επιλογή και 10% των νέων φαρμάκων παρουσιάζουν ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον κατά τους ισχυρισμούς των φαρμακευτικών ε, εταιριών. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις ανησυχίες. Συμπερασματικά θα ήθελα να αναφερθώ στις αμφιβολίες που κάποιοι μπορεί να έχουν στο θέμα της ενημέρωσης και της πληροφόρησης από πλευράς ασθενών. Υπάρχουν όμως ενώσεις ασθενών. Εγώ θα ήθελα να δω μία σχέση μεταξύ των κρατικών αρχών, των δημοσίων αρχών και των ασθενών. Παραδείγματος χάρη, τις τελευταίες αυτές ε, μέρες στη Γαλλία έχουμε εβδομάδες ευαισθητοποίησης και διαλόγου που οργανώνονται από τα μεγάλα φαρμακευτικά εργαστήρια, ούτως ώστε να ενημερωθούν οι οργανώσεις ασθενών πρόκειται κατά τη γνώμη μου για μια ενέργεια όπου η δημόσια αρχή ε, αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία για να ε, εξασφαλίσει μια ισορροπία ενημέρωσης. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά πάντως στη Γαλλία ε, συνέβη αυτό και με εξέπληξε που αυτή η εβδομάδα διαλόγου οργανώθηκε από μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία. Εξού και η ανάγκη για πρόσθετους ε, κανόνες όπως προτείνεται τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. <coughs> Κύριε Σταταρέλα. Presidente, io mi complimento con... Ε, ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια. Μας έδωσε μία, μας έκανε μία εκτεταμένη εισαγωγή εμπεριστατωμένη εισαγωγή και θα ήθελα μια εξήγηση είτε από την εισηγήτρια είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υπάρχουσα σχέση μεταξύ του συστήματος της Συγκεντρωτικής Τράπεζας Δεδομένων και των εθνικών κέντρων. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω πώς αυτά τα δύο θα ε, συνεργαστούν το Εθνικό Σύστημα και το Συγκεντρωτικό Κεντρικό Σύστημα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει σε ερωτήσεις σα. στο βαθμό που ήταν ερωτήσεις βέβαια. Παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κάρβεν και να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τις απόψεις που διατύπωσε, ε, περιλαμβανομένης και της συμβαστικής πρότασης η οποία ε, κατατίθεται. Θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια σχόλια των μελών αυτής της Επιτροπής και θα αρχίσω από την τελευταία παρέμβαση διότι είναι αρκετά σημαντικό για να αντιληφθούμε τα υπόλοιπα. Το κείμενο αυτό δεν μεταβάλλει την ευθύνη των χωρών μελών όσον αφορά την φαρμακοεπαγρύπνηση. Δεν υπάρχει μεταφορά ευθυνών από το εθνικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, παραδείγματο χάρη. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ε, ότι επιθυμούμε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο να συντονίζονται μεταξύ χωρών μελών και να υπάρχουν κοινέ αποφάσεις για την απόσυρση, τη μη απόσυρση, τη διαφοροποίηση των φαρμάκων κλπ. Διότι προς το παρόν έχουμε αποφάσεις εξατομικευμένες αν θέλετε ε, σε εθνικό επίπεδο ένα φάρμακο αποσύρεται σε μια χώρα δεν αποσύρεται σε μια άλλη κλπ. Εμείς λοιπόν επιθυμούμε να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των χωρών μελών. Ο ρόλος λοιπόν αυτής της βάσης δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης είναι να υπάρχει μια ενιαία βάση δεδομένων ε, προσβάσιμη, προσπελάσιμη από όλες τις εθνικές δημόσιες αρχές. Ωστόσο, οι αρμοδιότητες των εθνικών αρχών δεν μεταβάλλονται. Όσοι έχουν δικαίωμα να εισαγάγουν ε, ανεπιθύμητες ε, ε, αντιδράσεις ε, φαρμάκων είναι οι δημόσιες αρχές και τα φαρμακευτικά εργαστήρια. Ούτε εδώ λοιπόν υπάρχει αλλαγή. Όσον αφορά τον ασθενή, τους ασθενείς, το δικαίωμα των ασθενών. Να ενημερώνουν τις δημόσιες αρχές, δεν μεταβάλλεται. Αυτό λοιπόν που προβλέπουμε είναι οι ασθενείς να ενημερώνουν τις δημόσιες αρχές τους για μία ανεπιθύμητη ενέργεια, αντίδραση και οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να αξιολογήσουν αυτή την πληροφορία όπως αξιολογούν πληροφορίες που προέρχονται από γιατρούς, από νοσοκομεία ή από άλλες αρχές. Συνεπώς δεν υπάρχει ρήπανση σε εισαγωγικά των πληροφοριών με την ε, ενημέρωση από πλευράς ασθενών. Ε, ιδιαίτερως αυτές οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες για ε, φάρμακα τα οποία λαμβάνουν χωρίς ε, συνταγή. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να ενημερώσει ο ασθενής τις δημόσιες αρχές με τις συγκεκριμένες ε, πληροφορίες, υπάρχει ένας, ένα ολόκληρο πεδίο των φαρμακευτικών βιομηχανιών που δεν μπορούν να αξιολογήσουν αυτή την περίπτωση χωρίς ε, συνταγές. Το θέμα τώρα των φαρμάκων κοινόχρηστης ονομασίας. Και εκεί αυτά τα φάρμακα έχουν την ίδια υποχρέωση ε, ε, ενημέρωση σε περίπτωση ανεπιθύμινων αντιδράσεων. Τα φάρμακα κοινόχρηστης ε, ονομασίας είναι γνωστά φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά επί σειράν ετών και θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υποβάλουμε αυτά τα φάρμακα στο PSUR, δηλαδή στην περιοδική έκθεση ενημέρωσης ε, όπως συμβαίνει με τα νέα φάρμακα. Η κυρία Ριβαζή αναφέρθηκε στο ε, θέμα του ε, σχεδίου, του πλάνου αξιολόγησης της ε, κρίσης και τη σύγχυση που μπορεί να υπάρξει με την επιτήρηση ή εποπτεία της λειτουργίας του συστήματος. Είμαι πολύ σαφής. Η πρόταση αυτή δεν τροποποιεί, δεν μεταβάλλει τους κανόνες με τους οποίους η τα φάρμακα αξιολογούνται και μπαίνουν στην αγορά. Στην πρόταση αυτή δεν υπάρχει κανένα σημείο το οποίο να επηρεάζει ε, τον έλεγχο των φαρμάκων ε, πριν μπουν στην εμπορία, πριν διατεθούν στην εμπορία. Το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου είναι μια υποχρέωση επιπρόσθετη της φαρμακευτικής βιομηχανίας όταν, ε, ε, όταν ε, εμφανίζουν νέα καινοτόμα φάρμακα. Οι κλινικές δοκιμές ενδιαφέρουν έναν περιορισμένο πληθυσμό. Τώρα όσον αφορά στην διαφάνεια. Είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο με διάφορες προτάσεις, παραδείγματο χάρη θυμάμαι την, ε, τις προτάσεις για την παιδιατρική, ε, Όλες μας λοιπόν οι προτάσεις έχουν ως στόχο την μέγιστη δυνατή διαφάνεια, την ενημέρωση του κοινού για την ασφάλεια των φαρμάκων και για την έγκριση των φαρμάκων. Θεωρώ λοιπόν ότι στην πρόταση αυτή έχουμε μία σειρά διατάξεων που συνολικά δημιουργούν ένα ουσιαστικό σύστημα διαφάνειας. Δηλαδή δεν είναι μόνο το θέμα της πρόσβασης στην φαρμακοεπαγρύπνηση, διότι ε, στην, στην φαρμακοεπαγρύπνηση βεβαίως συγκεντρώνονται πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλά δεδομένα. Ωστόσο, ε, το να Γνωρίζουμε ότι στη Σουηδία είχαμε παραδείγματο χάρη ε, πέντε θανάτους εξαιτία ενό ε, εμβολίου χωρίς να γνωρίζουμε τις υπόλοιπε λεπτομέρειες. Αυτό είναι ανησυχητικό. Και αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ε, καταρχήν πρέπει να γνωρίζουμε αν αυτοί οι πέντε θάνατοι οφείλονται στον εμβολιασμό ή όχι. Και οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι στη διάθεση του κοινού, να μπορεί το κοινό να έχει πρόσβαση στις ε, πληροφορίες αυτές. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια μεγαλύτερη διαφάνεια, βεβαίως σεβόμενη ε, ε, την, τα προσωπικά δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επέστρεψε την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάνω στην πρόταση αυτή λέγοντας ότι το τελικό αποτέλεσμα η πρόταση η οποία θα εγκριθεί θα πρέπει να σέβεται την ανωνυμία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αναφέρεται το όνομα και τα προσωπικά δεδομένα στην ε, στα στοιχεία που δίδονται. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι και στις Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχουν αντίστοιχοι κανόνες με αυτήν της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, παραδείγματο χάρη, δεν είναι δυνατόν ένα Αμερικανό πολίτη ή ένα δικό μα πολίτη μέσα από εφημερίδε και από το ίντερνετ να εξασφαλίζει πληροφορίες, ενώ ο δικός μας ε, πολίτης δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Επίσης, θα ε, ε, προβλέπεται η οργάνωση δημοσίων ακροάσεων, ούτως ώστε αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν και να έχουν πληροφορίες από μια έρευνα η οποία έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές όπως ακριβώς και ε, στις πληροφορίες της Food and Drug Administration στις ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι πρόκειται για ένα επιπρόσθετο μέσο για να ενημερώνεται ο ασθενής για θέματα φαρμάκων και όπως πολλοί από εσάς επισημάνατε, οι οδηγίες που περιλαμβάνονται μέσα στα φάρμακα δεν είναι πάντοτε πάρα πολύ χρήσιμες και κατανοητές. Και πολλές φορές ο ασθενής παίρνει ένα φάρμακο χωρίς να έχει διαβάσει όλες τις οδηγίες. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό μία σύνοψη ε, των ε, πληροφοριών που ε, πληροφορίες τις οποίες έχει καταγράψει ο κατασκευαστής και που έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή να υπάρχουν πάνω στο ίδιο το φάρμακο. Νομίζω ότι απάντησα λίγο πολύ στις ερωτήσεις που μου υποβλήθηκαν, τις πιο σημαντικές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε τη Λίντα. Λίντα, θέλεις να πεις κάτι ακόμα? Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις αυτές. Ε, μπορείτε να μου στείλετε και γραπτός παρατηρήσεις. Δύο πράγματα να πω. Καταρχήν, ως προς τις ε, απευθείας αναφορές από τους ασθενείς. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να στείλουμε σε κάποιου συναδελφου κάποιε πληροφορίε για αυτό, διότι όπω είπε η Κομισιόν, δεν είναι ότι εγώ ω ασθενή έχω μια αντίδραση και μπορώ να βάλω τι πληροφορίε μου στην εθνική ή ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Ε, κανένας ασθενής δεν μπορεί να ε, βάλει πράγματα απευθεία στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Ε, απευθύνεται κανείς στην εθνική του αρχή και η αρχή αυτή, όπως κάνει και με τους γιατρούς και τους νοσοκόμους κτλ, εξετάζει τα στοιχεία και μπορεί να επανέλθει στον ασθενή, να απευθυνθεί στον ασθενή να ε, ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Και μόνο εφόσον εγκριθούν οι πληροφορίες αυτές από την Εθνική Αρχή προστίθενται στην βάση δεδομένων. Φοβάμαι ότι κάποιοι ασθενείς δεν ε, λένε πράγματα στο γιατρό τους, ε, παρότι ο γιατρός τους δίνει χρόνο για κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι κάποιοι μίλησαν για την άλλη πρόταση Φερχόγγεν, αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό θέμα, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Η δική μου θέση είναι ότι δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ε, απευθεία επαφή μεταξύ επιχειρήσεων, φαρμακευτικών εταιριών και ασθενών. Οι αρχές σε, τοπικό και, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο συλλέγουν τις πληροφορίες και αποφασίζουν τι θα τις κάνουν. Πρόκειται για τις ε, δημόσιες αρχές οι οποίες είναι κεντρικές στο σύστημα αυτό το θέμα εδώ πέρα αφορά τη δημόσια υγεία. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, όπως είναι άλλωστε και η διαφάνεια. Νομίζω ότι θα μπορούσα να συνδέσω κάποιες από τις, πληροφορίες, ε, κάποιες από τις παρατηρήσεις που έγιναν για το ε, για το φυλάδιο μέσα, στις, ε, μέσα στη συσκευασία ε, και ε, το θέμα της ενημέρωσης των ασθενών. Το θέμα δεν είναι ο μεγάλος όγκος πληροφοριών. Θα πρέπει οι παρενέργειες να αναφέρονται γραμμή προς γραμμή, μικρές και μεγάλες παρενέργειες. Εγώ αυτό που θέλω να ξέρω, αυτό που θέλω να ξέρει ο ασθενείς είναι μία σοβαρή ανάλυση που θα έχει γίνει από ανεξάρτητου ε, εμπειρογνώμονε ε, στη δημόσια υγεία. Νομίζω ότι αυτέ οι πληροφορίε θα πρέπει να διατίθεται στο κοινό και το ίδιο ισχύει για τα PSUR στα οποία αναφέρθηκε ο Πίτερ Λίζε. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσει στέλνουν αυτέ τι εκθέσει στι εθνικέ αρχέ. Νομίζω ότι μπορείτε να ρωτήσετε τι εθνικέ σα αρχέ τι τι κάνει τι εκθέσει αυτέ. Διότι πολλέ από αυτέ τι εκθέσει τη PSUR αποστέλλονται στι εθνικέ αρχέ, πολλέ από αυτέ ούτε καν τι ούτε καν τι διαβάζει κανεί διότι οι ε, εθνικές αρχές ε, έχουν υπερβολικό φόρτο, ε, υπερβολικό όγκο πληροφοριών. Θα πρέπει δηλαδή να εξαχθούν οι ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τα PSUR και αυτές να διαβιβάζονται. Όλες οι παρενέργειες αναφέρονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες και θα πρέπει οι εθνικές αρχές να μπορέσουν να συλλέξουν ε, θα πρέπει οι πληροφορίες αυτές να φιλτραριστούν για να συμπεριληφθούν στο PSUR και να σταλούν μετά στην Εθνική Αρχή. Υπάρχει ο κίνδυνος της πλημμύρας ε, των πληροφοριών, του κατακλυσμού πληροφοριών, Και υπάρχουν τόσε πληροφορίε στο ε, φυλάδιο που είναι μέσα στη συσκευασία ενός ε, ε, φαρμάκου που αν τα διαβάσω καταλαβαίνω ότι μπορεί να μου συμβεί οτιδήποτε αν πάρω το φάρμακο αυτό. Καλύτερα είναι να έχουμε κάποιες λίγες πληροφορίες κλειδιά ώστε ο ασθενής να ενημερώνεται σωστά. Κυρία Βιβάση, εγώ νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι φόρτος για τις επιχειρήσεις. Δεν τις διευκολύνει να διαθέσουν προϊόντα στην αγορά. Είναι άλλο ένα βήμα που πρέπει να κάνουν για τη δημόσια υγεία και κατά τη γνώμη μου ε, συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε ότι δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά ενό φαρμάκου. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους και προσλέπω στη συνέχιση τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε την έκθεση τη συνεδρία τη Επιτροπής το Γενάρη και ψηφοφορία ενδεχομένω στην Επιτροπή το Μάρτιο. Προετοιμαστείτε για αυτό το σημαντικό θέμα. Και πάμε στο 19 τώρα. Προφορική ερώτηση ε, της κυρίας Σου Σχετικά με προσωρινή αναστολή στα τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Η κυρία Γιούζο έχει το λόγο. Ή μήπως η μηπω η Επιτροπή για να απαντήσει απευθείας. Όπω θέλετε. Η κυρία Γιούσο πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε να απαντήσει Θέλω να κάνω κάποια προκαταρκτικά σχόλια. Νόμιζα ότι θα απαντούσε πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν πειράζει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πρέπει να σας πω καταρχάς ότι ανέλαβα ε, την υπόθεση αυτή ε, με τη νέα θητεία στο μέση, στα μέσα της διαδικασίας. Και ενώ οι πολιτικές ομάδες είχαν συμφωνήσει να αναβληθεί η κοινή θέση του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα μέχρι να οριστεί ο νέος Επίτροπος. Και να είμαστε βέβαιοι ότι όταν θα φτάσει στο Κοινοβούλιο κοινή θέση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να πάρει ε, αποφάσεις ε, με πολύ μεγαλύτερη νομιμοποίηση. Μπορεί αυτό να είναι σόφρον και προσεκτική απόφαση, αλλά ξέρετε ότι επήγει το θέμα, γιατί έχουμε νέες τεχνολογίες ε, την παραγωγή τροφίμων με κλωνοποιημένα ζώα και πρέπει εμείς να απαντήσουμε σε αυτό. Είναι ένας οικονομικός κλάδος που χρειάζεται καλύτερες απαντήσεις και νωρίτερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι τεχνικές ε, ε υποθέσεις. Χρειάζεται συζήτηση. Υπάρχουν θέματα δεοντολογίας, θέματα ευημερία των ζώων. Αλλά ε, υπάρχουν διάφορα επιχειρήματα τα οποία δεν ευσταθούν. Και κάθε ε, καταναλωτής μπορεί με τα λόγου γνώσεως ε, να αποφασίσει. Αν θέλει να αγοράσει ένα τρόφιμο που πρέχεται από ζώο κλωνοποιημένο, καλώς. Εμείς θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα τρόφιμα που κυκλοφορούν είναι ασφαλή και υγιεινά. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε κανένα καταναλωτή τα συναισθήματά μας, τις αποφάσεις μας, τις αντιλήψεις μας, γιατί δεν μπορούμε να κλωνοποιήσουμε την ανθρώπινη βούληση. Εγώ έτσι πιστεύω. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη ε, γενικά για το θέμα αυτό, ε, τουλάχιστον από τότε που το ανέλαβα. Λοιπόν, Αποφασίσαμε να το αναβάλουμε, αλλά ε, και μια που αναβλήθηκε είχα την ευκαιρία να συζητήσω και θα πρέπει να συζητήσουμε και εμείς να ενημερωθούμε, να δούμε ε, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα της πιθανής αναστολής, τη moratorium, Το συζητούν ε, οι ενδιαφερόμενοι να υπάρξει αναστολή, δικαιοστάσιο για τα τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Σας λέγω λοιπόν τι πιστεύω για το θέμα αυτό και τι προβλήματα μπορεί να προκαλέσει ε, αυτή η αναστολή ε, κυκλοφορίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πιστεύει από πλευράς νομικής. Ποιες θα ήταν οι συνέπειες αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο σε ό,τι αφορά την εισαγωγή ε, κλωνοποιημένων ζώων και τροφίμων πρώτης ή δεύτερης γενεάς από τρίτες χώρες πάντα και τα προβλήματα που μπορούμε να έχουμε, μπορούν να προκληθούν ε, στα πλαίσια του ΠΟΕ. Επίσης, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε περίπτωση που υπάρξει τέτοια απαγόρευση εισαγωγής τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα, πώς μπορεί να γίνει ένας επιστημονικός και τεχνικός έλεγχος. Ένα κλωνοποιημένο ζώο, εντάξει, είναι κλωνοποιημένο το ζώο. Εάν ε, είναι ο πατέρας του κλωνοποιημένος ή το δικό του παιδί ή το, το, ζώο που θα γεννήσει το κλωνοποιημένο. Πώς θα καταλάβω εγώ ότι είναι κλωνοποιημένο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Στην Ισπανία ε, υπάρχει ε, ένα ε, σταύρος σε ένα εκτροφείο πολύ υψηλής ποιότητας για αναπαραγωγή χρησιμοποιείται και για τη σπερματέγχυση δεν θα το σφάξουν το ζώο είναι πάρα πολύ καλό για τις σταυρομαχίες και παράγονται ταύροι και έχουν κάνουν και ουρά ε, ε, μετά και στα κρεοπολία ε, για να αγοράσουν κρέας αυτού του ταύρου μετά την ταυρομαχία. Και είναι σίγουρο ότι θα γεμίσουν τα κρεοπολία της Ισπανίας από γόνους αυτού του ταύρου που είναι κλωνοποιημένος και έχει γίνει χαμός στην Ισπανία. Αυτό όλο ποιος θα τα ελέγξει. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσει κανείς την προέλευση. Ο Παόλο Τεστόρη, ε, αναπληρωτής διευθυντής ε, από την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, θα μας δώσει πληροφορίες. Παρακαλώ. Η κυρία Παόλα Σαρτόρη, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Αγιούζο που έθεσε την ερώτηση αυτή που μας επιτρέπει να διευκρινίσουμε το πολύ δύσκολο αυτό ζήτημα. ζήτημα. Πριν απαντήσω, θα ήθελα να πω και να επιβεβαιώσω ότι η Επιτροπή ήδη έχει κάνει βήματα απαραίτητα για να διασφαλιστεί η κάλυψη οποιοδήποτε κινδύνου για τον χρήστη από την κλωνοποίηση. Και να σας πω και γιατί, διότι το 2008 όταν προέκυψε αυτό το θέμα της κλωνοποίηση. ζητήσαμε από την ΕΦΣΑ να γνωμοδοτήσει ε, όσον αφορά το κρέας από κλωνοποιημένα ζώα. Και η ΕΦΣΑ μας είπε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την ασφάλεια τροφίμων ε, ανάμεσα ε, σε ζώα κλωνοποιημένα σε σχέση με τα συμβατικά ζώα. Η ΕΦΣΑ το 2008 είπε ότι όπως και να έχει υπάρχει έλλειψη στοιχείων και γνώσης και ότι χρειάζεται περισσο... περαιτέρω έρευνα. Φέτος ζητήσαμε από την ΕΦΣΑ να εξετάσει τα νέα επιστημονικά στοιχεία και μας επιβεβαίωσε ότι σύμφωνα με αυτά δεν υπάρχει καμία διαφορά όσον αφορά την ασφάλεια. Τι καλύπτει ήδη η νομοθεσία μας. Ήδη έχουμε νομοθεσία που καλύπτει την πώληση προϊόντων και την ε, υγεία των ζώων. Η νομοθεσία αυτή λέει ότι όλα τα ζώα, ακόμα και αν είναι κλωνοποιημένα, θα πρέπει να ε, πληρούν τα κριτήρια και να ε, και να μπορεί να εντοπιστεί η προέλευσή τους, να είναι ανοιχνεύσιμα. Επίσης ε, δεν ε, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι που να ε, βλάπτουν τα ζώα και όσον αφορά τα τρόφιμα, ο παρόν κανονισμός για τα νέα τρόφιμα, τα novel foods, καλύπτει το, τα τρόφιμα από ζώα. ακόμα δηλαδή και αν δεν τροποποιήσουμε την ομοθεσία, καλύπτονται τα τρόφιμα από ζώα όσον αφορά την έγκριση πριν τη διάθεση στην αγορά. Διασφαλίζεται λοιπόν ένα επίπεδο προστασίας. Να απαντήσω στην ε, κυρία Αγιούζο. Ποιες θα είναι οι συνέπειες ε, σε σχέση με τις διεθνείς συμφωνίες. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθετήσει για τα κλωνοποιημένα ζώα θα πρέπει ε, η νομοθεσία να συνάδει με τον ΠΟΕ. Τρεις συμφωνίες του ΠΟΕ μπορεί να μας ενδιαφέρουν εδώ. Καταρχήν, η λεγόμενη συμφωνία SPS που καλύπτει όλα τα μέτρα ε, που έχουν να κάνουν με την ε, υγειονομική προστασία. Εάν θέλουμε να αιτιολογήσουμε έναν περιορισμό στο εμπόριο στα πλαίσια του SPS, θα πρέπει να υπάρχει κίνδυνος από τη χρήση του προϊόντος αυτού. Και όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή η ΕΦΣΑ δεν ε, θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος για την ε, ασφάλεια. Θα είναι δύσκολο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αιτιολογήσει μέτρα στα πλαίσια του SPS. Θα μπορούσαμε βέβαια πάντα να λάβουμε προσωρινά μέτρα και με βάση την αρχή της προφύλαξης, διότι πάντα υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε περίπτωση αβεβαιότητας. Πιστεύουμε όμως ότι θα είναι πολύ δύσκολο να υπερασπιστούμε τέτοια μέτρα σε επίπεδο ε, ΠΟΕ. Ο δεύτερο τύπο μέτρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα DBT, τα η τεχνική φραγμή στο εμπόριο. Θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε υποχρέωση επισήμανση. Υπάρχουν όμω και εδώ κανόνε. Δηλαδή, εάν εφαρμόσουμε τέτοια μέτρα, θα πρέπει να το αιτιολογήσουμε αυτό με βάση το δικαίωμα του καταναλωτή να, για ενημέρωση θα πρέπει να δείξουμε ότι στην Ευρώπη ο καταναλωτής θέλει, και εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε το δικαίωμα του αυτό, να γνωρίζει από πού προέρχεται το προϊόν. Έχουμε τα ευρωβαρόμετρα. Τα φετινά ευρωβαρόμετρα μας λένε ότι ο Ευρωπαίος καταναλωτής θέλει να γνωρίζει. Η τρίτη συμφωνία στα πλαίσια του ε, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι η συμφωνία GATT που μας επιτρέπει να λάβουμε μέτρα που είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουμε ε, το, το κοινό. Το άρθρο 20 της Συμφωνίας ΓΚΑΤ επιτρέπει τέτοια μέτρα. Ωστόσο, θα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο μη αυθαίρετο και δεν θα πρέπει να πρόκειται για καλυμμένη καλυμμένο περιορισμό στο διεθνές εμπόριο. Θα πρέπει δηλαδή να λάβουμε υπόψη την αρχή της αναλογικότητας. Κλείνοντας, ε, ως προς το πρώτο ερώτημα, να πω ότι Ελλείψει σαφούς κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία ή την υγεία των ζώων, ο περιορισμός ε, στην πώληση ε, προϊόντων από κλωνοποιημένα ζώα θα ήταν δύσκολο να σταθεί. ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής από τρίτη χώρα. Δεύτερη ερώτηση. Τι δυνατότητα υπάρχει να ελεγχθεί η κίνηση η διακίνηση των ε, προϊόντων από κλωνοποιημένα ζώα. Συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει τρόπος διάκρισης των τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα και από συμβατικά ζώα. Τα τρόφιμα είναι όμοια. Εάν επιβάλλουμε απαγόρευση θα πρέπει να επιβάλλουμε και μέτρα ανιχνευσιμότητας του ζώου και του τροφίμου, διότι το ίδιο το, το προϊόν δεν διαφέρει. Θα πρέπει δηλαδή να ανιχνεύσουμε την πορεία του ζώου για να γνωρίζουμε εάν το προϊόν προέρχεται από κλωνοποιημένο ζώο ή από ε, απόγονο κλωνοποιημένου ζώου. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε μέτρα ανιχνευσιμότητας εκτός της Ευρώπης, διότι δεν μπορεί ε, η νομοθεσία μας να είναι εξωεδαφική. Θα πρέπει λοιπόν να επιβάλλουμε σε όλες τις εισαγωγές ένα σύστημα ε, πιστοποιητικών, τα οποία θα πρέπει να είναι επίσημα, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι το προϊόν αυτό δεν προέρχεται ούτε από κλωνοποιημένα ζώα, ούτε από απογόνους τους. Ελπίζω να σας έδωσε κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι οριστικά. Όπως σας είπα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα τα θέματα αυτά. Αλλά μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι η Κομισιόν συνεχίζει να εξετάζει όλες τις στοιχείες της κλωνοποίησης ε, και το νέο σώμα των επιτρόπων θα ξαναεξετάσει το ζήτημα αυτό κατά τη δεύτερη ανάγνωση του κανονισμού για τα νέα τρόφιμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τεστόρη. Πολύ λίγο χρόνο έχουμε. Θα παρακαλούσα τους αδέρφους να μιλήσουν δύο λεπτά ο καθένας. Ο κύριος Λίζε είναι πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Γιούζο για την ερώτηση αυτή και ευχαριστώ την κυρία Τεστόρη που απάντησε. Ωστόσο, θα πρέπει να επαναφέρω την ισορροπία. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στις διάφορες πολιτικές ομάδες. Ε, όταν ε, το συζητήθηκε το θέμα, ασχολήθηκε και το ΕΛΚ με το θέμα αυτό. Με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ζητήσαμε απαγόρευση και μάλιστα γενική απαγόρευση. Ξέρω ότι υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες. Δεν το αρνούμε αυτό. Οι παρατηρήσεις της κυρίας Τεστόρη όμως ήταν κάπως ελλειπείς. Υπάρχει γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ, πράγματι. Υπάρχει όμως ε, και ε, γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Ηθικής, EGE, e, όπου υπάρχουν ε, ισχυρά επιχειρήματα υπέρ μιας απαγόρευσης. Η προστασία των ζώων αποτελεί, μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα στον ΠΟΕ, διότι τα, τα ζώα που κλωνοποιούνται υποφέρουν. Θα πρέπει, πιστεύω, να εξετάσουμε δηλαδή περαιτέρω το θέμα της διάθεσης στην αγορά του κρέατος ε, των ε, απογόνων των κλωροποιημένων ζώων. Θα πρέπει να καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες. Εάν δεν κάνω πολύ λάθος όμως, το θέμα είναι και η επισήμανση. Εάν θέλουμε να έχουμε επισήμανση στα ζώα, ε, στους απογόνους κλωνοποιημένων ζώων, αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσανατολιστούμε σύμφωνα με την έκθεση Λιωτάρ και την ε, θέση του Νίλ Πάρης. Το να απεμπολίσουμε τη θέση όμως του Κοινοβουλίου βρίσκω ότι είναι πολύ πρόημο αυτή τη στιγμή. Να εξετάσουμε λοιπόν την, τη γνωμοδότηση του EGE ε, και ε, τα, τα άλλα σχετικά κείμενα, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε σχετικά μέτρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πέτερ Λίζε. Να ρωτήσουμε την κυρία Τεστόρη εάν ε, ελήφθη υπόψη η προστασία των ζώων κατά, την, κατά τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ η Ευρώπη. Θέλει στον ΠΟΕ να υπερασπιστεί την προστασία των ζώων. Αυτό δεν αναγνωρίζεται ακόμα όμως στα πλαίσια του ΠΟΕ. Αυτή είναι η διαπραγματευτική μας θέση. Εάν είναι να ληφθεί ένα μέτρο που να βασίζεται αποκλειστικά στην ε, ευζοία των ζώων, την προστασία του, του, του συμφέροντος του ζώου, αυτό θα είναι δύσκολο να γίνει στα πλαίσια του ΠΟΕ. Ευχαριστώ. Ωραία. Η κυρία Σάπο για το θέμα αυτό, παρακαλώ. Vreau uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα και εγώ της προφορικής ερώτησης και του δικαιοστασίου και το θέμα της επιμερίας των ζώων, αλλά με κάλυψαν οι συνάδελφοι, οπότε θα ήθελα να πω το εξή εγώ μόνο. Άκουσα ότι ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ξέρει τι καταναλώνει υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι καλά ενημερωμένος. Και εμείς πώς θα εγγυηθούμε ότι οι ε, πληροφορίες που μας δίνει ο παραγωγός είναι σωστές. Και πώς μπορεί να ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα εισαγόμενα προϊόντα προέρχονται ή δεν προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Αυτό πώς ελέγχεται, πώς επαληθεύεται. Γιατί έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα ήδη με αυτά τα θέματα. Φοβάμαι ότι είναι σχεδόν αδύνατο να το ελέγξουμε. Μιλώ για τα εισαγόμενα πάντα προϊόντα. Και αφού ανοίξουμε αυτούς τους ασκούς, δεν πρόκειται τίποτα να ελέγξουμε από εκεί και πέρα. Μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έχουν πρόβλημα τα κλωνοποιημένα τρόφιμα, αλλά να το ξέρουμε. Μπορεί ο άλλος να θέλει να τα αγοράσει, αλλά ξέρει τι αγοράζει. Ερώτηση της κυρίας Κάτεμπαχ. Τεχνικά υπάρχει δυνατότητα να λέμε στη σήμανση το αντίστροφο, ότι σε αυτό το προϊόν δεν καταφέραμε να ανοιχνεύσουμε την προέλευσή του. Και να το λέει επάνω, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αυτό ρωτάω. Να μην λέμε προέλευση τάδε, απλώς αγνώστου προελεύσεως. Η κυρία Τεστόρη. Thank you Ευχαριστώ. Όπως ανέφερα στην απάντησή μου, η σαφή σήμανση είναι εφικτή. Η σήμανση θα πρέπει να βασίζεται στην πλήρη ανεχνευσιμότητα του ζώου. Ε, δηλαδή να ξέρουμε την προέλευση, ότι είναι κλόνος, ότι χρησιμοποιήθηκε για λόγους αναπαραγωγής, και ότι γεννήθηκαν δεκάδες, εκατοντάδες ε, άλλα ζώα κλπ. Μπορεί κανείς να εφαρμόσει ένα σύστημα ανιχνευσιμότητας, ε, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί και επίσης πάρα πολύ βαρύ, δύσκολο από διοικητική σκοπιάς. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε στην Ευρώπη γιατί έχουμε πλήρη ανιχνευσιμότητα στις χώρες μέλη των ζώων. Ήδη εφαρμόζεται ένα τέτοιο σύστημα από τη στιγμή που γεννιέται ένα ε, ζώο, έχει ένα διαβατήριο με όλες τις πληροφορίες. Για τις εισαγωγές θα πρέπει να υποχρεώσουμε τις τρίτες χώρες να εφαρμόσουν ένα σύστημα ανιχνευσιμότητας το οποίο κάποιες χώρες δεν έχουν. Θα μπορούσαμε και θα πρέπει να το δικαιολογήσουμε στο ε, με δυσκολίες. Εν πάση περιπτώσει όμως το νόημα είναι πολύ δύσκολος ο έλεγχος, ε, δαπανηρός. Όλα είναι εφικτά. Δεν λέω ότι δεν είναι εφικτό, αλλά πρέπει κανείς ε, να αναλογιστεί και την αναλογικότητα. Και η κυρία Βίζια που αναφέρθηκε στην, στο κώδικα ηθικής και την Ευρωπαϊκή Ομάδα, κώδικα δεοντολογίας, ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο του, της ε, ΓΚΑΤ, δηλαδή το ηθικό συμφέρον ή το ε, ε, ηθική προστασία, αν, θέλα, θέλετε. Ωστόσο, δεν είναι τόσο ξεκάθαρη και οριστική όταν λένε ότι μάλλον δεν ζητούν μια, μια απόλυτη απαγόρευση με την αναστολή της ε, λειτουργίας. Ιδιαίτερα όταν αναφέρονται ε, το, στον κλόνο και στους ε, προγόνους του κλόνου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λίζε δέχτηκε μια απάντηση, δεν σας άκουγε, αλλά θα του το διαβιβάσουμε αυτά που είπατε. όχι, δεν θα ξανακάνει την ερώτηση την άλλη φορά που θα το συζητήσουμε, γιατί του απαντήσανε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τελειώνει η συζήτηση για το σημείο 19 και ερχόμαστε στο 20 σύντομα απολογισμό της επίσκεψης της αντιπροσωπείας στην Ουάσιγκτον. Έχουμε μια σύντομη έκθεση. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πολύ συναρπαστική η αποστολή εκεί της αντιπροσωπείας μας. Ευχαριστώ και τη γραμματεία. Είχαμε πολλές επαφές στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ε, στη Γερουσία, ε, με την κυβέρνηση, ε, με την οικονομία, με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ε, αποκομίσαμε μια εικόνα λοιπόν, πλήρη νομίζω για την κατάσταση των συζητήσεων εκεί. Ξέρετε ότι έχει γίνει μεγάλη αλλαγή από την κυβέρνηση Μπού στην κυβέρνηση Ομπάμα. Δεν χωράει καμία αμφιβολία φαίνεται ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι και ε, σωστό και είναι ότι έχουν επιστρέψει πλέον οι Ηνωμένε Πολιτείε σε αυτή τη διαδικασία, την νομοθετική, όλα αυτά τα μέτρα για την προστασία από την κλιματική αλλαγή. Και το θέμα είναι τι θα γίνει μέχρι την Κοπεχάγη τώρα και τη διάσκεψη που έχουμε σε λίγες εβδομάδες το πιθανότερο είναι ότι δεν πρόκειται να γίνουν και πολλά ακόμα, διότι η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση στο σύστημα υγείας είναι υπαριθμόν ένα προτεραιότητα. Και δεύτερη ε, είναι η υπόθεση της καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής. Οπότε εκκρεμεί ακόμα αυτό το θέμα της Κοπεχάγης. Δεν ξέρουμε αν οι Αμερικανοί θα φέρουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, αν μπορούν, ε, είναι σε θέση ωστόσο. Δεν είναι σίγουρο καν αν θα έρθει ο ίδιος ο Ομπάμα στην Κοπενχάγη. Όλα αυτά είναι πολύ θολά και αόριστα και συγκεχημένα και αν είναι έτσι πολύ βασανιστική κατάσταση μάλλον δεν θα έρθει. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν παρόμοια συστήματα στη συζήτηση ε, και θέματα τους απασχολούν όπως και εμάς. Οι ε, ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας, το σύστημα εκπομπών και σαν το ETS κάτι που λέγεται cap and trade περίπου τι συζητήσει κάνουν για τα ενεργειακά και αυτά που συζητάμε κι εμείς. Είναι μεγάλη πρόκληση να περάσει ένας νόμος από τη Γερουσία, γιατί χρειάζεται 60 ψήφους από τις 100 και ενδεχομένως να γίνονται συμβιβασμοί που δεν είναι πάρα πολύ ε, χρήσιμοι, ούτε απαιτούνται για το κλίμα, οι γερουσιαστές αγωνίζονται σκληρά και μάχονται τα λόμπι για ε, την πολιτεία του ο καθένας. Από τη μια έχει στον άθρακα που η χαλιβουργία ε, ε, είναι τεράστια βιομηχανία, η πετρελαιοβιομηχανία, βιομηχανία, ξέρετε ότι δίνονται περισσότερες άδειες από ό,τι έχουν προβλεφθεί ως τώρα για γεωτρήσεις, offshore, μπροστά στις ακτές, προνόμια στον άνθρακα, στην πυρηνική ενέργεια και στις διερευνητικές ε, γεωτρήσεις για φυσικό αέριο. Οπότε πού να χωρέσουν οι καημένοι σε ανανεώσιμες εκεί μέσα, όταν έχουμε τόσα πολλά ενεργειακά λόμπι ε, που ε, διαγωνίζονται. Ελπίζουμε λοιπόν στην Κοπεχάγη να συναντηθούμε με πολλούς εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει μεγάλη δέσμευση, προσήλωση των ε, βουλευτών που θέλουν να γίνουν ε, προσπάθειες και πρόοδοι. Θα προσπαθήσουμε στην Κοπεχάγη να ε, διοργανώσουμε και κοινέ δραστηριότητες. Και πέρα από την Κοπεχάγη, αυτή η σχέση και η συνεργασία Ευρώπης-Αμερικής είναι υπαρξιακή σημασία για την υπόθεση της κλιματικής αλλαγής και είμαστε αισιόδοξοι. Το επόμενο διάστημα μπορούν να εμφανιστούν σημαντικέ πρόοδοι και στι ΗΠΑ. Ευχαριστώ όλα τα μέλη που ήρθαν στην αντιπροσωπεία. Το πρόγραμμα ήταν πολύ ελκυστικό, ενδιαφέρον, αλλά και πάρα πολύ βαρύ. Από νωρί το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Άξιζε τον κόπο που πήγαμε εκεί. Τώρα ξέρουμε περισσότερα και μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα με τι ΗΠΑ. Αυτά. Όσα αναφορά εισαγωγικά για την αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον, η κυρία Ντεμπρούνα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω μαζί σας για να ευχαριστήσω τη Γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Πράγματι είχαμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα και πολύ καλές συναντήσεις, ενημερώσεις και άλλες συνεδριάσεις προετοιμασίας. Η Γραμματεία έκανε εξαιρετική δουλειά. Συμφωνώ ότι είχαμε μια πολύ καλή και ενδιαφέρουσα σειρά συναντήσεων όχι μόνο στο Κογκρέσο από τους ε, κυρίους και κυρίες γερουσιαστές, αλλά επίσης και στο Υπουργείο Ενέργειας και επίσης με προσώπους πολύ σημαντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο ήταν η συζήτηση με το US CAP στην οποία συμμετέχουν ε, πέντε μεγάλες ε, ΜΚΟ και ε, καμιά δεκαπαντεριά μεγάλες εταιρείες οι οποίες οι οποίοι όλοι μαζί θέλουν να υπάρξει μια ειδική νομοθεσία για το περιβάλλον. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ ενδιαφέρον, μπορούμε να συνεργαστούμε να, για να επηρεάσουμε θετικά, θετικά την νομοθεσία. Επίσης, όπως είπε και ο πρόεδρος, είναι αυτή η αίσθηση της νέας προσέγγισης. Αν κάποιος είχε πάει προηγουμένως στην Ουάσιγκτον πέρσι, παραδείγματος χάρη, και από την προσωρινή Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή ήταν απολύτως σαφές ε, για αυτόν που ξέρει και το παρελθόν ότι υπάρχει μια εντελώς νέα προσέγγιση με την κυβέρνηση Ομπάμα σε σχέση με την κυβέρνηση Μπούς. Ε, από την άλλη βεβαίω υπάρχουν όλα αυτά τα σύνθετα προβλήματα ε, στι ΗΠΑ και μπορεί να μην καταλήξουμε στην γι' αυτό είναι προφανές. Εν πάση περιπτώσει, ε, Εμεί θέλουμε να έχουμε τις μέγιστες δυνατέ συναντήσεις με τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω τι ευελιξία έχουμε ε, για το ταξίδι, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τα μεγέθη των άλλων αντιπροσωπιών και ε, επίσης με τα δύο μέλη της γραμματείας που ήταν μαζί μας στις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα ήταν χρήσιμο να είναι μαζί μας στην Κοπεχάγη, ακριβώς για να κυνηγήσουν, λέει η κυρία, τους ανθρώπους με τους οποίους συναντηθήκαμε στις Ηνωμένε Πολιτείες και να έχουμε επαφή μαζί τους. Δεν ξέρω πώς μπορεί να καλυφθεί αυτό. Επίσης, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε ενημέρωση, πληροφόρηση σε καθημερινή βάση. Είχαμε κάποιες πληροφορίες μετά την επιστροφή μας, αλλά είναι χρήσιμο να συνεχίσουμε να ενημερωνόμαστε για χρηματοδοτήσεις από την κυβέρνηση Ομπάμα σε διάφορες πρωτοβουλίες. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως όλες οι βιομηχανικές χώρες θα πρέπει να επιδείξουν με μεγαλύτερες, μεγαλύτερη φιλοδοξία για να επιτευχθεί ο στόχος που έχουμε θέσει. Ευχαριστώ. Είναι ε, και 25 έτσι, πάει πίσω το ρολόι. Προσοχή, ο Κρήτον Αρσένης, παρακαλώ. Thank you very much. I will speak in Greek. Ε, πραγματικά θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για την εξαιρετική δουλειά που έγινε. Ε, πολύ γρήγορα, απλά να αφαιρθώ ότι πραγματικά είναι εντυπωσιακή η αλλαγή της τάσης της, ε, στην Αμερική, τον είπα, με την, μετά την εκλογή του Προέδρου Ομπάμα. Παρόλα αυτά ε, και φαίνεται και η εκτίμησή μου είναι ότι τελικά στο τέλος της, ε, όλης αυτής της περίοδου είτε μέσω νομοθεσίας είτε μέσω ρύθμισης, regulation, θα έχουμε τελικά ε, μειώσεις, μια πολιτική μειώση των ακουμπών του θερμοκηπίου αντίστοιχη αυτή της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελικά. Παρ' όλα αυτά, ε, πραγματικά είναι πολύ αβέβαιη η στάση της Αμερικής στην Κοπεχάγη και θα είναι πολύ δύσκολο και η επικύρωση μιας απόφασης ε, από, την, ε, από τη Γερουσία. Γι' αυτό πραγματικά θα πρέπει όλοι μας να ανεβάζουμε όσο είναι δυνατόν τους, τον παλμό ε, τον, να υπεθυμίζουμε στην Αμερική ε, ότι υπάρχει ένα πολιτικό κόστος από το να μην είναι μέρος μιας διεθνής συμφωνίας. Δεν φτάνει μόνο να κάνει τη δικιά της δουλειά άψογα και σωστά που πιστεύω θα την κάνει. Ε, είναι πολύ σημαντικό να δεσμεύσουμε όλα τα μέρη του πλανήτη σε μια διεθνή δεσμευτική συμφωνία με μετρήσιμους ποσοτικούς στόχους. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς, αυτός είναι ο στόχος. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναδούμε μέχρι την Κοπενχάγη. Θα τα ξαναπούμε. Θα δούμε τι εφόδια θα έχουμε και πώς θα διοργανώσουμε αυτές τις συναντήσεις με τους άλλους. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Η δουλειά συνεχίζεται και μετά την Κοπενχάγη και θα πρέπει να διατηρούμε στενές επαφές με την Αμερικανική πλευρά. Σας ευχαριστώ πολύ και τους διερμηνείς. Καλωσύνη σας. Λήξεις μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Στο καλό να πάτε.